Just So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, 9 και 7 λεπτά πήγε και όλοι διαμαρτύρονται ότι δεν μας φτάνει η ώρα. η μόνη δυνατότητα να έχουμε χρόνο είναι να ξεκινάμε γκέρος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Σκάιερ, τον Γενικό Εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2017. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 10, συζήτηση για το Γενικό Προϋπολογισμό του 2017. Χθες κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Είχαμε μία επιστολή από τον ε, κύριο και τον εισηγητή μας, την ψηφίσαμε, η οποία επιστολή περιείχε τις ε, προτεραιότητες της εντολής για τον τριμερή διάλογο. Έτσι ώστε να έχουμε τη δική μας ε, θέση και το τι επιθυμούμε. Το 2017, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα έτος με πολλά στοιχεία που μας αφορούν με τη στρατηγική εμπόριο για όλους, το Trade for All, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Διαπραγματεύσεις με την Κίνα, με χώρες της Ασίας, με τις χώρες ΑΚΕ, Μεξικό, Χιλή, και με τον εξυγχρονισμό των ε, σχετικών συμφωνιών. Επίσης, έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία ΤΙΖΑ και πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα του ΠΟΕ, πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε και να εξετάσουμε όλες τις πτυχές, που είναι αρκετά πολλές. Ε, έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε ως προς το νομοθετικό μας έργο. Και φυσικά αυτό έχει και οικονομικές πτυχές. Στην στρατηγική εμπόριο για όλους έχουν προσθεθεί και κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Για παράδειγμα, ανταγωνιστικό ένας διαγωνισμός για τις ε, πόλεις fair trade στην Ευρώπη πρέπει να διοργανωθεί. Επίσης κάτι άλλο το οποίο θεωρώ αρκετά σημαντικό. δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τις διαπραγματεύσεις, αλλά και με την εφαρμογή. Και η εφαρμογή, εφαρμογή πρέπει να στηριχθεί οικονομικά. Με τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε τι έχουμε καταφέρει και αν το δούμε αυτό τότε θα αρχίσουμε να κουνάμε το κεφάλι μας, διότι στην εφαρμογή δεν έχουν γίνει αυτά που προσδοκούμε. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέρυσι για πρώτη φορά έγιναν περικοπές στο προσωπικό της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Και φυσικά δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι η εμπορική πολιτική είναι το μέσο για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι το ουσιαστικό, το, το μέσος που εφαρμόζουμε την εξωτερική μας πολιτική στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν, Γιάννης, έχουμε μεγάλες απαιτήσεις για το τι περιμένουμε από τον προϋπολογισμό του 2017. Για το τι θέλουμε να δούμε στον προϋπολογισμό, για το ποιες είναι οι αρμοδιότητες και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις προτεραιότητες στην πράξη. Ήρθες εδώ για να μας καθησυχάσεις, ελπίζω, για να μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι το βράδυ, γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες μας θα εκπληρωθούν. Γι' αυτό λοιπόν σου δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά Μπέρντ. 24 Μαΐου έχουμε σήμερα. Πριν από μερικές εβδομάδες Ήμουν αρκετά ανήσυχος. Είχα άγχος για αυτή τη μέρα, διότι αυτή η μέρα ήταν εκείνη όπου θα μας παρουσίαζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προϋπολογισμό του 2017. Αυτό για μένα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι άλλαξαν τα πάντα στη ροή των εργασιών μου, στην καθημερινότητά μου και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα περί τα τέλη του 2017, έτσι ώστε να μπορέσω να εκπληρώσω το έργο μου. Τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε την παρουσίαση του προϋπολογισμού και οι πληροφορίες μου λένε ότι η αναβολή αυτή θα είναι για τέσσερις εβδομάδες, περίπου δηλαδή στις 26 και 27 Ιουνίου. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει τίποτα με τις 23 Ιουνίου, με το Συμβούλιο δηλαδή, αλλά πιο πολύ από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, τα, με το πρόσθετο κόστος για την προσφυγική κρίση, ότι δεν έχουν κάνει καλά τον υπολογισμό και ότι έχουν προκύψει νέες ανάγκες. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί τόσο αυτή η εξήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επειδή ακόμα δεν γνωρίζω τι έχουν κατά νου, μπορώ να κάνω κάποιες εικασίες σχετικά με το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της απόφασης για αναβολή. Και θα μπορούσα να κάνω μερικές εικασίες σχετικά με τις επιθυμίες ή με τις ε, προσδοκίες μας. Πιστεύω πάντως πως στο τέλος θα καταφέρουμε να δώσουμε μία λύση. Πιστεύω πως το Κοινοβούλιο θα καταφέρει να ενωθεί πίσω από μια κοινή θέση ως προς τον προϋπολογισμό. Όμως να ξέρετε πως δεν είμαστε μόνοι μας στις διαπραγματεύσεις και επίσης και δυστυχώς δεν είμαστε στην ευχάριστη θέση που είχαμε πριν τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Αυτό θεωρώ πως είναι ένα μειονέκτημα από τη... που έχει προκύψει από τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Πρέπει να συμφωνήσουμε με την Προεδρία του Συμβουλίου η οποία αυτή τη στιγμή έχει μία σύνθεση η οποία ελάχιστα έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, η Επίτροπος Γεωργίευα, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, τα έχει περιγράψει έτσι με πολύ ωραίο γλαφυρό τρόπο. Μας έχει πει ότι το Συμβούλιο δηλαδή έχει χωριστεί στα τρία. Έχει τρία μέτωπα. Το μέτωπο της γεωργίας, το μέτωπο της συνοχής και το μέτωπο των εκπτώσεων. Τώρα για το που ανήκει η χώρα μου, πιστεύω πως δεν χρειάζεται να το πω. Το Συμβούλιο τι κάνει λοιπόν. Προσπαθεί μαζί με μας να κατέβει μια κοινή θέση. Όμως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γλιτώσουν χρήματα. Και επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Τον Απρίλιο, κατά την συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, συζητήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές τις δικές μας για τον προϋπολογισμό του 2017. Τις ψηφίσαμε, τις υπερψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία. Γι' αυτό λοιπόν αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση και μεγάλη ευχαρίστηση που καταφέραμε να είμαστε τόσο πολύ ενωμένοι. Είναι όμως δύσκολα τα πράγματα και περίπλοκα. Κατά τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον τωρινό προϋπολογισμό του 2016, τα περιθώρια σε σημαντικές κατηγορίες του προϋπολογισμού έχουν αλλάξει. Δηλαδή, κατηγορία 3, περιβαλλοντική πολιτική, και στην κατηγορία 4, στην εξωτερική πολιτική, έχουν γίνει λοιπόν αλλαγές και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα περιθώρια που έχουμε μέχρι τέλους εξαιτίας ακριβώς της ε, προσφυγικής κρίσης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει πολλά ειδικά μέσα τα οποία διαθέτουμε στην, στο πλωστάσιό μας τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα διότι πρόκειται για ειδικά μέσα, μέσα ευελιξίας του προϋπολογισμού, τα οποία είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Δηλαδή, χωρίς την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα ως προς την απόφαση, θα ήταν πιο εύκολα. Τώρα, έχουμε αρκετό περιθώριο ελιγμών, από τη μία, για τον προϋπολογισμό, Καταφέραμε να επηρεάσουμε τον προϋπολογισμό του 2016, όμως δεν έχουμε δει ακόμα τις αλλαγές φέτος. Και αυτό οφείλεται σε πολλά. Αυτό οφείλεται στην κατάσταση στη Συρία, όπου οδήγησε εκατομμύρια πολίτες στην προσφυγιά. Από την... Και είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να συνυπολογιστεί αυτό το κόστος στον προϋπολογισμό. Αυτό μας απασχόλησε για τον προϋπολογισμό του 2016. Κινητοποιήσαμε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ και πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Επίσης, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη. Χρειάζεται τόνωση μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μετά, στο πολιτικό περιβάλλον. 3,38 δισεκατομμύρια πρέπει να κινητοποιηθούν για, την... για τις εγγύησεις του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν και εδώ να προσθεθούν αυτά τα κονδύλια στον προϋπολογισμό. και η πολιτική κατάσταση έχει ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του χρόνου θα ε, περιμένει εμάς να τοποθετηθούμε πάνω στην μεταρρύθμιση και στην αναθεώρηση, με συγχωρείτε, του προϋπολογισμού. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα, το σε δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι όπως ήταν. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο λιτότητας και η πίεση γι' αυτό οφείλεται στη δική μου κυβέρνηση. Όμως αυτή η πίεση είχε ασκηθεί προτού η Ευρώπη μπει σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, προτού αρχίσει να υφίσταται τέτοιες έντονες πιέσεις. Μετά, Πρέπει να αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να συνδεθεί με τον προϋπολογισμό. Έχουμε τα διάφορα έγγραφα που μας έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη ε, της Ευρώπης. Έχουμε τις ετήσιες εκθέσεις για την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όλα αυτά μας δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Συνεπώς λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στον προϋπολογισμό εξαιτία όλων αυτών. Χρειάζεται βελτίωση λοιπόν. Επίσης υπάρχουν και πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες έχουν ζητηθεί από εμάς. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της φτώχειας, η ενίσχυση ε, των νέων, της νεανικής επιχειρηματικότητας, ε, η στρατηγική 2020. Αυτά είναι σημεία που δεν πρέπει να ξεχνάμε και που πρέπει να ενισχύσουμε. Επίσης, Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβάλει την ε, δημοσίευση της πρότασής της. Τώρα, εμείς πρέπει να αποχωριστούμε το εξής. Πρέπει να αποχωριστούμε δηλαδή την ε, επιθυμία μας να συμμετέχουμε με εντολή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δηλαδή, η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα συμπεριληφθεί ως παράρτημα στις γενικότερες συστάσεις. Αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2014, στον προπολογισμό του 2014, όταν βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο και δεν είχαμε καθόλου χρόνο ή ελάχιστο έστω χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε με το Συμβούλιο να συζητήσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διατυπώσουμε τη δική μας. Εμείς δηλαδή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχάς θα εργαστούμε με τις συστάσεις του Συμβουλίου και όχι με δικές μας. Δηλαδή όχι, δεν θα τοποθετηθούμε άμεσα. Δεν θα ασχοληθούμε άμεσα με το κείμενο της Επιτροπής, αλλά με τις ε, προτάσεις και συστάσεις του Συμβουλίου πάνω σε αυτό το έγγραφο της Επιτροπής. Σε γενικές γραμμές αυτό που διαβάζω είναι οικονομία, εξοικονόμηση πόρων, ελαχιστοποίηση δαπανών. Και βλέπω πως στη συζήτηση στο Συμβούλιο κυριεύει το θέμα της εφαρμογής. Δηλαδή, έτσι όπως έχει τοποθετηθεί το Συμβούλιο, μέσω των εθνικών οικονομικών αρχών, βλέπω ότι δεν έχει εστιάσει τόσο στο περιεχόμενο. Βλέπουν όμως τους ρυθμούς, ε, ε, τα ποσοστά εφαρμογής. Δεν κοιτάζουν την ουσία. Και εκεί μας λένε ότι ναι, αν δεν εφαρμοστεί το πρόγραμμα σημαίνει ότι δεν λειτουργεί και αν δεν λειτουργεί τότε, τότε δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσα κονδύλια, τότε μπορούμε να κάνουμε περικοπές και να γλιτώσουμε λεφτά. Χωρίς όμως να, γνωρί... να φαίνεται γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί κάτι δεν λειτουργεί. Εγώ προσπαθώ να εμποδίσω να γίνει κάτι τέτοιο, να γίνουν περικοπές, όμως βλέπω ότι η εφαρμογή για το 2015 τουλάχιστον δεν είχε καλά ποσοστά επιτυχίας, άρα δεν νομίζω να γίνει κάτι. Νομίζω μάλιστα πως θα γίνει αυτό που φοβάμαι. Σίγουρα δεν έχουμε έναν προϋπολογισμό γενναιόδωρο και μάλλον βλέπω ότι αυτό που γίνεται είναι πως ε, περνάνε με τη θεριστική μηχανή και κόβουν-κόβουν. έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση. Το Συμβούλιο δηλαδή εξαιτία της ε, μη ικανοποιητική εφαρμογή να κάνει περικοπέ, να επέμβει και να κάνει περικοπέ. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτά ήταν λοιπόν τα αρχικά μου σχόλια, προσπαθώντα να σας παρουσιάσω το πλαίσιο και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα βλέπω πως δεν μας δίνεις και πολλές ελπίδες, έτσι να το πω χοντρά. Τι λέει ο συγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Γέννης, μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπες. Όμως πιστεύω πως ίσως έχουμε κάνει ένα λάθος στις τελικές διαπραγματεύσεις του πολιτισμού νομικού πλαισίου. στο τελικό στάδιο βλέπουμε ότι τα ανώτερα όρια πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία. Υπάρχει μια κατανομή, όμως χρειάζεται να συμφωνήσουμε για αυτήν την ευελιξία. Χωρίς την ευελιξία αυτή που είναι αναγκαία δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ταυτόχρονα τι βλέπω. Βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει τεράστια δημιουργικότητα στα σχέδιά της, δηλαδή έχει προτείνει πράγματα τα οποία μας προσπερνούν και ταυτόχρονα απορώ με αυτά που προτείνουν. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης και πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και όλες τις εναλλακτικέ λύσεις που έχουμε, έτσι ώστε να καταρτήσουμε έναν σωστό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα που αφορούν τη δική μας Επιτροπή, τα προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Γειτονία, για παράδειγμα, δεν θέλει να δει τα προγράμματα μας, θέλει ε, να δει τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε. Δεν θέλει να δει δηλαδή την εφαρμογή στην πράξη. Θέλει να τις ε, πούμε πώς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα σταθεροποιήσουμε την ε, κατάσταση στη γειτονία, γειτονία μας. Αυτό λοιπόν φαίνεται πως παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το 2017 αλλά και για το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα ασχοληθούμε όχι μόνο με ε, τα οικονομικά αλλά με το στρατηγικό σχεδιασμό. Πώς δηλαδή θα πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που θέλουμε με τα μέσα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω. Μετά, με το Ταμείο για την... Ε, Βόρεια Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπω ότι κάνει απελπισμένες προσπάθειες να παρακάμψει αυτήν την αναθεώρηση με την δικαιολογία ότι μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα αναθέτοντάς το εξωτερικά παρά συζητώντα το εδώ. Προσπαθεί δηλαδή να παρακάμψει τις υφιστάμενες δομές. και να παρακάμψει δηλαδή το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλές φορές, για παράδειγμα λέει, ωραία, εάν ας πούμε το κράτος, ε, κάθε κράτος μέλος συνεισφέρει 3 δισεκατομμύρια, τότε εντάξει, δεν χρειάζεται ε, να το συζητήσουμε παραπέρα. Έχουμε το ταμείο μας για... και δεν ξέρω όμως αν λειτουργεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει επιτυχία ένα τέτοιο πλάνο. Προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει κάτι τέτοιο, για μένα θα πρέπει να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα συνηγορήσουμε σε μια τέτοια πρόταση. Διότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ποια είναι τα όρια μα. Επίση, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα πώ συνδέεται ο προπολογισμό του 2017 με την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε σαφείς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περισσότερο από ποτέ πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός περισσότερο ε, βασισμένος στις θέσεις του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μετά από όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γένς είχε δίκιο όταν μας ανέφερε τους λόγους για τους ε, οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβάλει την παρουσίαση του προϋπολογισμού. Για αυτές τις δυσκολίες που μόλις αναφέρθηκαν. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Μογκερίνη ε, προτίθεται να δημιουργήσουν νέα ταμεία, νέες προτάσεις που ε, που θα είναι, που θα έχουν 60, μέχρι 60 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργία διάφορων ταμείων και πολλά από αυτά τα κονδύλια θα ε, ταμεία θα χρησιμοποιήσουν κονδύλια από άλλα ταμεία, από τα διαρθρωτικά ταμεία για παράδειγμα. Είναι κάτι που παρουσιάστηκε πρώτη φορά πριν από μερικές εβδομάδες. Πώς πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που έχουμε, πρόσθετες δυνατότητες. Τώρα, η κυρία Μοκερίνη και ο κύριος Τίμερμανς θέλουν να μας παρουσιάσουν αυτό το νέο σχέδιο αρχές Ιουνίου. Και ελπίζουν να ε, εγκριθεί το σχέδιο αυτό πριν την ε, σύνοδο του Ιουνίου 2018. Στη σύνοδο του στις 28 Ιουνίου. Δηλαδή τι θα γίνει τότε, το Συμβούλιο θα αποφασίσει κάτι και εμείς απλά θα το δεχτούμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει ε, δεν θα νομοθετήσει. Εσείς τι λέτε να κάνουμε με αυτά που ακούσατε, λέτε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι το Συμβούλιο πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το ότι αν δεν μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση, γιατί σε κρίση βρισκόμαστε, αν δεν αρχίσει να, ε, αν δεν αρχίσει να... αν δεν αναγνωρίσει μάλλον το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί η κρίση, πρέπει να αφήσει τα πράγματα να γίνουν σύμφωνα με την ε, συνήθινη νομοθετική διαδικασία. Και αυτή συμπεριλαμβάνει εμάς. Πρέπει να γίνει ανταλλαγή απόψεων, πρέπει να ακουστεί η δική μας άποψη η άποψη των αρμόδιων επιτροπών και να γίνει αυτό τον Ιούνιο. Πρέπει να, να καταβάλουμε λοιπόν προσπάθειες για να το κάνουμε αυτό και να μην περιμένουμε τι θα γίνει, να μην έρθουμε ούτε εμείς ούτε το Συμβούλιο πρώτο Τελεσμένου Γεγονότος. Ε, τώρα, κύριε Πρόεδρε, ίσως δεν είναι απόλυτα σχετικό με αυτά που λέμε, αλλά θα το αναφέρω γιατί πιστεύω ότι μας αφορά. Ψηφίσαμε μια πρόταση αρκετά αμφιλεγόμενη. Για το... Ψηφίσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων το 2016 ε, όσον αφορά το εμπόριο. Ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο και στην ε, δημιουργία του αλλά και στα επόμενα στάδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι, δεν, ότι αυτό έχει να κάνει με αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι δεν συμφωνούμε με αυτό. Θα πρέπει να αναλύσουμε την πρόταση αυτή για να δούμε αν είναι σωστό ή όχι. Βλέπω όμως ότι Αυτές οι αποφάσεις σχετικά με την ε, συνδιαλλαγή, αυτό που είχαμε προτείνει δηλαδή εμείς, δεν υπάρχουν. Έχουν βγει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι χειραγώγηση του χείριστου του είδους. Δεν είναι μία μικρότητα, κάτι ασήμαντο. Εδώ είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Και περιμένω από εσάς μέχρι το καλοκαίρι να έχετε ε, διορθώσει το λάθος. Ε, περιμένω την αρμόδια επίτροπο να δηλώσει δημόσια ότι θα διορθωθεί και γυρίζω και το λέω σε εσά. Διότι να ξέρετε ότι αυτό δείχνει μεγάλη αλαζονία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακάμπτει έτσι το Κοινοβούλιο. Ντροπή σας! Και όταν γίνονται τέτοια πράγματα σε, τόσο, ε, σε τέτοια προγράμματα, φανταστείτε τι έχει να γίνει και σε πιο σοβαρά θέματα. Άσχετα με το τι άποψη έχει ο καθένα για τον προπολογισμό, όταν, όταν λαμβάνεται μία απόφαση, αυτή πρέπει να εφαρμόζεται. Και αναμένω και εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεση απάντηση για το τι έχει γίνει και πώ ε, προτίθεται να το διορθώσει. Αυτά λοιπόν. Τώρα, χθε με τους ε, συντονιστέ. αποφασίσαμε για τα βασικά σημεία στα οποία θα στηριχτούμε για την διαδικασία του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις αντίστοιχες ε, τροπολογίες. Εδώ πιστεύω πως η τεχνική στήριξη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αλλά υπάρχει και η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τεχνική στήριξη στα πλαίσια των, του, της διαδικασίας προϋπολογισμού, δηλαδή στήριξη όπου παρατηρούνται αδυναμίες διοικητικού τύπου. τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή διοικητικά των ε, μέσων του προπολογισμού. Αλλά αυτό πιστεύω πως χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τονίζει αυτό, σε κάθε ευκαιρία, ότι δεν θέλει να κάνουμε μικροδιαχείριση, δεν θέλει να παρεμβαίνουμε στις δικές της αρμοδιότητες, αλλά εδώ αναφέρονται περικοπές στο, προ... στο προσωπικό, επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών στις διάφορες γενικές διευθύνσεις, εξακολουθητικός ε, έλεγχος, όμως βλέπω ότι όλα αυτά έχουν πολλές ε, παγίδες. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, διότι αφορούν πολλούς τομείς, όχι μόνο για παράδειγμα τη συμφωνία TTIP, αλλά και άλλα. Χρειάζεται λοιπόν εμείς να κάνουμε τις αναλύσεις μας να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλες τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Μετά, υπάρχει και το θέμα της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά αυτήν εδώ την Επιτροπή άμεσα. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στις ε, πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Σούστερ έχει το λόγο από το S&D. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω αρχικά με όσα έχουν υποθεί. Δεν βρίσκομαι πολύ καιρό σε αυτή την επιτροπή έτσι ώστε να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες του προπολογισμού. Όμως βλέπω ότι πράγματι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ε, εφαρμόσει τι κατευθυντήριε γραμμέ που μα αφορούν. Τώρα, θα αναφερθώ σε ένα σημείο γιατί δεν θέλω να επαναλάβω όσα έχουν υποθεί, αλλά το θεωρώ σημαντικό. Ο κύριος Μπόγκε μας είπε για αυτές τις ε, αποφάσεις που λαμβάνει το ε, Συμβούλιο, λες και είναι ε, παντοδύναμο. Ορισμένα από τα ταμεία στα οποία αναφέρθηκε έχουν συσταθεί γιατί υπήρξε ανάγκη. Σίγουρα υπάρχουν αμφιβολίες, αλλά πιστεύω πως, όπως είπε και ο Λάνια και ο κύριος Μπέγκε, εάν θέλουμε να πάρουμε την εμπορική μας στρατηγική στα σοβαρά, πιστεύω πως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα τα οποία θα, έχουν, θα δώσουν προστιθέμενη αξία, θα έχουν θετικά αποτελέσματα και πώς θα εφαρμοστούν αλλά και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά έξω, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά δεν πρέπει να αφήσουμε το θέμα αυτό μόνο σε, στα χέρια τεχνοκρατών και εμπειρογνωμόνων, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε ευρύτερο πλαίσιο με την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Και αυτό εμείς ως πολιτικοί έχουμε υποχρέωση να το εξασφαλίσουμε προτού ολοκληρωθούν οι εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά, να, να δούμε την συνέχεια και να είναι μια συνέχεια η οποία θα μας ικανοποιεί. Αυτό λοιπόν θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ε, στα πλαίσια των διαφυλάξεων για τον προπολογισμό. Τι θα γίνει δηλαδή στο μέλλον και μάλιστα ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι έρχεται μια δύσκολη αμφιλεγόμενη συμφωνία, συμφωνία σύνδεση, ε, εταιρικής σχέσης με τις αφρικανικές χώρες. Προτού λοιπόν υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να παραμερίσουμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν προσφυγικά ρεύματα που φεύγουν από αυτές τις χώρες. Πρέπει να δούμε το γενικότερο πολιτικό ε, πλαίσιο προτού καταφύγουμε στα διάφορα ταμεία έκτακτης ανάγκης, βοηθητικά ταμεία κτλ. Και σίγουρα χρειάζεται, πιστεύω, να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευελιξία την οποία αναφέρουμε. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν τη μεγάλη σημασία που έχει όχι μόνο αυτή η εμπορική συμφωνία, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο πίσω από αυτή και οι επιπτώσεις μετά από αυτή. Η εφαρμογή δηλαδή και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Αυτά με τις ε, επιθυμίες αυτές της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Λάμπστορφ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού, αλλά με αυτά που ακούω θα, θα αρχίσω τα αντικαταθλιπτικά. Ο προϋπολογισμός δηλαδή έχει αναβληθεί εξαιτία του Brexit για να έχουμε δηλαδή χρόνο να συζητήσουμε για την εντολή, να συζητήσουμε για το πολιτέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας αναφέρει θέματα ευελιξίας έτσι ώστε να ακολουθήσει τους δικούς της ε, στόχους. Και δεν ξέρω πραγματικά με αυτές τις ε, τοποθετήσεις, με περικοπές μάλιστα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα επιτύχει τους στόχους ε, που θέλει. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις έχω. Καταρχάς, αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τι θεωρεί πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία σε αυτό. Έπειτα, MFA, διαγραφή των MFA, τι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις. Μετά, οι αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ημινομοθετικό χαρακτήρα, είναι πολύ σημαντικές. Μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου μέσου. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και πιστεύω πως χρειάζονται γενικά εξηγήσει γιατί έχουμε απορίες. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου τη ΓΚΟΕ ο κύριος Σόλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πολύ μίζερα τα βλέπω τα πράγματα, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητέ για την παρουσίασή τους. Πιστεύω πως όντως πρέπει να προβληματιστούμε για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία που αφορούν αυτήν την Επιτροπή και να σας εκθέσω τις δικές μας απόψεις. Καταρχάς, πιστεύω πως έχουμε αυξημένες... Ε, έχουν αυξηθεί εμπορικές συμφωνίες και έχει αναφερθεί επίσης η επανεισαγωγή δασμών. Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει την εσωτερική αγορά και δεν διαθέτουμε άλλα κονδύλια πέρα από αυτό. Τώρα, Πώ θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ίδιου πόρου ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα κατά τις ε, διαβουλεύσεις. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να συνεισφέρει το κάθε κράτος μέλος στον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική και μια στρατηγική σε περίπτωση που δεν ε, λειτουργήσει η προηγούμενη στρατηγική και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό στα χέρια της Επιτροπής. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ και πιστεύω πρέπει να προβληματιστούμε άλλοι. Τώρα, στο καταστατικό αναφέρεται ότι το 2% του ΑΕΠ των κρατών μελών θα πρέπει να ε, δίνεται προς, προς το ΝΑΤΟ. Αυτό πιστεύω πως πρέπει να αναλογιστούμε εάν είναι λογικό. Εάν ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό και γενικότερα να επανεξετάσουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Σίγουρα θα μπορούσαμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα, ε, θα προσκρούσει πάνω στις συνθήκες και το πρόβλημα θα διαιωνιστεί. Τι γίνεται, φέρνουμε γύρω-γύρω το πρόβλημα, δεν δίνουμε όμως λύση. Μετά, συμφωνώ με τον κύριο Μπέγκε απόλυτα με το ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εμάς για αυτήν την ε, ευελιξία. Πρέπει αυτή η ευελιξία να μην γίνει σε βάρος άλλων σημαντικότερων υποχρεώσεων. Από τη μία δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να δεχτούμε ε, αυξημένο αριθμό ανθρώπων από άλλες χώρες, και από την άλλη όμως να μην βοηθάμε, τη, να μην δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε αυτές τις χώρες έτσι ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και από την άλλη ε, πρέπει επίσης να συζητήσουμε το θέμα της ε, συνεργασίας με αυτές τις χώρες. Ε, με αυτές Τι γίνεται με τα κριτήρια τα περιβαλλοντικά, με τα κριτήρια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να, πρέπει να εργαστούμε πάνω, στο, πάνω στην εξάλληψη των αιτίων που δημιουργούν ανάγκη και ανέχεια στις ε, τρίτες χώρες. Και πρέπει να καταστεί σαφές ότι χρειάζεται μια αλλαγή της ε, πολιτικής μας προσέγγισης. Και αυτό να φαίνεται και στον, ε, και στον προϋπολογισμό και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε λεπτά το πολύ. Κυρία Άλπατραν, Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση μόλις έγινε για ένα θέμα που δεν σχετίζεται μόνο με εμπορικά ζητήματα αλλά και υπερβαίνει και τις αρμοδιότητες αν θέλετε της Επιτροπής αλλά και της γενικής μας διεύθυνσης. Οπότε θα προσπαθήσω εγώ τώρα να ε, προσφέρω μία απάντηση στις παρατηρήσεις που κάνατε, οι οποίες όμως σχετίζονται με την εμπορική πολιτική. Είναι ξεκάθαρο πως ε, δεν είναι το πλέον θετικό, το γενικότερο πλαίσιο του προϋπολογισμού και το τόνισε αυτό επαρκώς ο εισηγητής. Και ως εκ τούτου έχουν ανακύψει δυσκολίες, ε, μεταξύ άλλων και για την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο το προσχέδιο. Δυστυχώς δεν έχω πιο συγκεκριμένη απάντηση για το πότε θα είναι διαθέσιμο. Φαίνεται από τα σχόλιά σας επίσης πως γενικότερα υποστηρίζετε ε, τους στόχους μας ως προς την εμπορική πολιτική, εκλαμβάνεται δε το εμπόριο ως ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε μεταξύ άλλων και το μεταναστευτικό ε, στις γειτονικέ μας χώρες αλλά και στην Αφρική οι δράσεις μας ακριβώς αυτό αποσκοπούν. Φυσικά έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολίων που αντιμετωπίζουμε λόγω ανεπαρκούς κατανομής κονδυλίων. Ε, διαρκώς εξελίσσεται το θεματολόγιο μας πολλοί άριθμους πρωτοβουλίες ε, προκύπτουν από την ανακοίνωση Trade for All για όλους από τον Οκτώβριο δηλαδή του 2015 και η παρακολούθηση και η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών που έχουμε διαπραγματευτεί έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, ε, όχι μόνο από τον Οκτώβριο πέρυσι αλλά και νωρίτερα. Ο επιχειρησιακό προπολογισμό τη ΓΔ Εμπορίου, και το θυμίζω είναι μικρό, ε, διοχετεύεται ω επιτοπλίστων σε αυτέ τι δραστηριότητε, δηλαδή η αξιολόγηση των συμφωνιών και σε διάφορες άλλες ενέργειες που στόχο έχουν την αύξηση της διαφάνειας για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής, δηλαδή συναντήσεις με τους φορείς της των πολιτών ε, τις ε, διοργανώνουμε συστηματικά όχι μόνο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ε, γιατί έχουμε πέρα από τις μελέτες της αξιολόγησης αντικτύπου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προβλέπονται συστηματικά τέτοιες συναντήσεις. Ε, σημείωσα τις παρατηρήσεις των βουλευτών μεταξύ άλλων και για τα πιλωτικά προγράμματα. Έχουμε ένα εξάλλου που σχετίζεται με ένα από τα θέματα που σχολιάσατε, δηλαδή τη διαφάνεια για την TTIP, Εξεργαζόμαστε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και θα σε ενημερώσουμε σύντομα για τις εξελίξεις. Αναφερθήκατε στην ε, κατάργηση αυτού του προγράμματος από, τα από τον κατάλογο των πιλωτικών προγραμμάτων και ο λόγος είναι ότι εγγραφεί σε μια γραμμή προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στις διοικητικές δαπάνες. Ε, δυστυχώς τα σχόλια του κυρίου Μπέγκη γίνονται εκτός μικροφών. Απάντησε. Στο παρελθόν ε, σας ε, το έχω πει και ε, συνεχώς απευθύνουμε έκκληση προς για να βρούμε ένα τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δραστηριότητες μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό το πρόγραμμα καθίσταται αδύνατο διότι το περιεχόμενο του, επειδή είναι επιχειρησιακό το πρόγραμμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη γραμμή που αντιστοιχεί στι διοικητικέ δαπάνε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι όμω είμαστε στη διάθεσή σα να το συζητήσουμε και μετά την συνεδρίαση μπορούμε να συνεχίσουμε διμερώς αυτή τη συζήτηση. Αυτό το πρόγραμμα είναι προς συμφέρον όλων και ε, καλύπτει τη χρηματοδότηση των μη για τα εμπορικά ζητήματα και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους. Δεν έχουμε κάτι εναντίον του ε, προγράμματος ε, και ε, εμπίπτει πλήρως στο πλαίσιο της εμπορικής μας πολιτικής. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσει για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν τελικά να συμπεριληφθούν στο θεματολόγιο δράσεων της ΔΕΛΤΑ Trade. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, γενικότερες όμως ερωτήσεις και ειδικότερε για αυτό το πρόγραμμα γέννηση είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Μια παρατήρηση για τον εισηγητή μας, αλλά και θέλω να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο πρόσωπος της Επιτροπής δεν έχει να κάνει μόνο με το αν το, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Έχει να κάνει με τη διαδικασία συνδιαλλαγή και με τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν αναμένω από την Επιτροπή και να, ε, να μας εξηγήσει γιατί έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ και γιατί και έχει κάνει το αντίθετο από τις αποφάσεις που έχει λάβει από εμάς. Μετά, βλέπω ότι έχουν γίνει συμφωνίες για ε, συμφωνίες όπως για παράδειγμα εκείνη του Λονδίνου, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει δηλαδή κάποιες ε, αποφάσεις τις οποίες δεν έχει εφαρμόσει. Και εμείς εδώ πρέπει να ε, αναπτύξουμε ένα νέο σύστημα για τον προπολογισμό που να δίνει περισσότερη διαφάνεια και ταυτόχρονα, ε, πέρα από το συζήτηση που κάνουμε εδώ, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο ε, για ε, τα διεθνή ταμεία έκτακτης ανάγκης, διεθνή ταμεία βοήθειας, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών και διαπιστώνω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε εάν είμαστε σε θέση αυτές τις μακροπρόθεσμες προοπτικές να τις εφαρμόσουμε εγκαίρως. Αν, δω αν δείτε δηλαδή τα νούμερα για το 2014 και 2015, θα δούμε ότι το 2015 είχαμε λιγότερα μέσα από ότι το 2014, παρότι ε, επιδεινώθηκε η κρίση. Και οι ε, μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις των συμμετεχόντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, μειωθεί. Πώς μπορούμε τώρα εμείς ε, να τις ε, συμπεριλάβουμε, ε, να, να τις αγκυροβολήσουμε στον προπολογισμό, έτσι ώστε κανείς στο μέλλον να μην μας κατηγορήσει ότι δεν ε, εκπληρώνουμε, ότι, δεν τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γένς. Τώρα θα σου δώσω λοιπόν ε, για το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα τα χρειαστώ τα πέντε λεπτά. αλλά θα ήθελα να σταθώ σε, ορισμένες, σε ορισμένα σχόλια. Καταρχάς, ε, τα σχόλια του κυρίου Λάμστορφ μας είπε για την ε, μακροοικονομική βοήθεια και ότι τα ποσοστά εφαρμογής δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε. Το Συμβούλιο τι κάνει, ε, κοιτάζει Κοιτάζει τα ποσοστά λοιπόν απορρόφησης και βλέπει εάν αυτά δικαιολογούν περικοπές ή όχι. Όταν παρατηρεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε παίρνει ένα κόκκινο μολύβι και σβήνει, διαγράφει. Δεν πιστεύω βέβαια να γίνει κάτι τέτοιο στην πράξη, όμως ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, να δούμε ίσως ξανά τα κείμενα. Τώρα, ε, να ευχαριστήσω πολύ τον Ράιμερ Μπέογκε. Πολλά από αυτά που είπε είναι ε, πολύ σημαντικά και ειδικά για αυτήν εδώ την Επιτροπή. Όμως, ε, να σταθώ σε συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχάς, για τα καταπιστεύματα, για τα trust funds. Χρειάζεται μία τακτική και ενδελεχής ε, εξέταση των πραγμάτων. Έχουμε καταρχάς ε, την νομοθεσία που μας επιτρέπει την δημιουργία καταπιστευμάτων, διότι είναι απόρρια της ε, ιδέας που είχαμε να ενώσουμε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για ένα κοινό σκοπό. Τι γίνεται όμως τώρα, τι έχουμε δει. Καταρχάς ότι ο έλεγχος των κονδυλίων, η διακυβέρνηση και το είπες ξεκάθαρα, Ράιμερ, έχει φύγει από τα χέρια μας στην ουσία. Και δεύτερον, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ γρήγορα κατάφερε να διαθέσει τα κονδύλια αυτά και δεν έχουμε δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις ε, αποφάσεις. Μας έφυγαν κονδύλια στο, ε, σε τελική ανάλυση. Έπειτα το είπες ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών είναι συμβολικές, δεν είναι ουσιαστικές και πραγματικά προκύπτει το ερώτημα ότι αν δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά αυτό το μέσο, γιατί το χρησιμοποιούμε, γιατί το δημιουργήσαμε. Και έπειτα βλέπουμε πως ε, υπάρχουν και, μικρά, και μικρό ποσοστό απορρόφησης. Τώρα, στο επόμενο καταπίστευμα που θα δημιουργηθεί, εμείς θα έπρεπε να πούμε ότι ναι, είμαστε σε θέση να συζητήσουμε, αλλά υπό ορισμένε προϋποθέσεις. Και ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον για το τρέχον έτος να αλλάξουμε τα πράγματα και να αφαιρέσουμε τη δική μας ε, συμμετοχή εφόσον δεν μετρά ο λόγος μας. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει πράγματι, υπάρχουν πράγματι τρύπε στον προπολογισμό και προσπαθούμε να τι μπαλώσουμε παίρνοντα κονδύλια από ένα ταμείο και βάζοντα τα σε άλλο. Αλλά αυτό δημιουργεί άλλε τρύπε. Σίγουρα δεν είναι σοβαρό τρόπο άσκηση πολιτική αυτό. Έπειτα, ο κύριος Λάμστορφ μας ε, είπε πως πρέπει να δούμε ποιε είναι, ποιες είναι οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Οι προτεραιότητες είναι αυτές που ακούσαμε. Σίγουρα αυτή η έκθεση καθιστά σαφές ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει υποστεί περικοπές. Είναι μικρότερο από ότι το προηγούμενο. Παρότι έχει επιδεινωθεί η κρίση και έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες. Αυτό μπορούμε φυσικά να το αφήσουμε χωρίς αντίδραση, αλλά θα δούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν και μεγάλη προθυμία να αλλάξουν τα πράγματα, διότι δεν έχουν τι να πούν στους πολίτες τους. Και μάλιστα οι αναγκαίες αποφάσεις είναι, δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στα κράτη-μέλη. Μετά, η έκθεση αναφέρεται και στους ίδιους πόρους και μη με παρεξηγείτε, και εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, αλλά αυτό συνεπάγεται και αφαίρεση ιδίων πόρων. Ήδη οι πόροι δημιουργούνται ε, από τους ε, δασμούς και εάν καταργηθούν οι δασμοί, μειώνονται και ήδη οι πόροι. Σας το λέω έτσι πολύ χοντρά. Αυτό δηλαδή δημιουργεί και ένα νέο ερώτημα. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα σύστημα ίδιων πόρων το οποίο θα στηρίζεται σε εισφορές ε, ποσοστού του ΑΕΠ από τα κράτη-μέλη. Κανείς δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Και να είστε σίγουροι ότι εάν ε, διατυπωθεί μια τέτοια πρόταση, τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να διαφωνούν και θα αρχίσει το ένα να κατηγορεί το άλλο κτλ. Θα υπάρχουν σίγουρα διαφωνίε σχετικά με τι προτεραιότητε που θα έχει το κάθε κράτο μέλο, προτεραιότητε χρηματοδότηση και σίγουρα δεν θα καταφέρουμε τίποτα με αυτό. Τώρα, εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τον προπολογισμό, πρέπει να έχουμε καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Πρέπει να επανεξετάσουμε τις κατηγορίες και να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συζήτηση και τις προτάσεις και τα σχόλιά σας. Πρέπει να φύγω δυστυχώ τώρα γιατί θα ε, πρέπει να πάω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όμως είμαι στην διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Σκάιερ που ήρθε εδώ και μας παρουσίασε αυτή τη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Τώρα, το επόμενο σημείο θα το αναβάλουμε για μετά την ψηφοφορία, το σημείο 11, και περνάμε αμέσω στο σημείο 12. Όπω ξέρετε, πρέπει να έχετε μαζί σα τι κάρτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα κάνουμε μια δοκιμή τώρα. Ελπίζω να έχετε όλοι τις ε, κάρτες. άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Jeder abgestimmt. Ψηφίσατε. Dann schließe ich die Testabstimmung. Ε, την πέραση της δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Ωραία, περνάμε στο σημείο 12. Τότε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τινησία. Πρώτη τροπολογία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 απορρίπτεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Ευχαριστώ, η κυρία Σάντζας. Σαρνέζ, συγγνώμη. Και τώρα σημείο 13. Αναθεώρηση συμφωνίας της Γενέβης για τα οχήματα και την τυποποίηση. Μόνο μία ψηφοφορία έχουμε. Άρχεται. Πέρας. Συντριπτική πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Τέλεια. Παρακάτω. 14. Ε, η Συμφωνία για την Τεχνολογία των Πληροφοριών. Και εδώ μία μόνο ψηφοφορία έχουμε. Άρχεται. Πέρας. Επίσης με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Σημείο 15 προφορική ερώτηση για τις επιπτώσεις ε, των κυρώσεων των ΙΠΑ στο Ιράν για τις επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχεται. Πέρας. Με μεγάλη πλειοψηφία επίσης εγκρίνεται και άρα θα υποβληθεί από την Επιτροπή μας στη συνέχεια και περνάμε στο σημείο 16 γνωμοδότηση για το νομικό πλαίσιο για τις ε, παραβιάσεις ε, το, της θελωνιακής νομοθεσίας και σχετικές κυρώσεις. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, ξέχασα την τροπολογία 2. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Γιατί 2 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τη συμβαστική την ψηφίσαμε, την συμβαστική 1 και περνάμε στο σημείο 4, τροπολογία μάλλον 4, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 23 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να γίνει μια επαλήθευση για την 24 παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παρακαλώ ε, σε να σκόντε τα χέρια για να ψηφίζετε. 28 ε, τώρα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 ε, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 32 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 33 τώρα. και εδώ είναι σε δύο τμήματα η ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα για την ε, τοπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 33 με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Τώρα, 35 σε δύο τμήματα επίσης. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα γίνει επαλήθευση και για αυτή. Για το πρώτο τμήμα της 35, παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται η 10 υπέρ κατά. Απόχες εγκρίνεται η 36 υπέρ κατά. Απόχες εγκρίνεται η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 12 με την προφορική τροπολογία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα έχουμε την ε, ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία άρχεται πέρας Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε, συγχαρητήρια και τώρα ε, σημείο 17 προετοιμασία της ε, αναθεώρησης του Πουδουπού ε, τροπολογίες 4 ε, και 5 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 1 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές Επαλήθευση παρακαλώ για την ε, τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίθηκε η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη, τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τώρα 12 υπέρ. Ορίστε. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Ε, θέλετε ελεγχό. Για τη 12. Ωραία, επαλήθευση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για τη 14 άρχεται πέρας απορρίπτεται η 15 και η 16 μαζί υπέρ όχι, λάθος λέει ο πρόεδρος, ε, επειδή έχουμε τη συμβαστική, ε, καταπίπτει. Mm. 18 και 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 28 και 29 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 37 υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε μια επαλήθευση για τη 37 άρχεται πέρας απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται. Πέρας. Επίσης με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αυτά για, την, ε, για τις ψηφοφορίες ολοκληρώνεται ο γύρος και περνάμε, ε, γυρνάμε πίσω μας στο σημείο 11 για τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών, μελών, των κρατών ΣΟΕΣ. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι, αν κάποιος θέλει να αποχωρήσει από την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνει με ησυχία. Σας παρακαλώ ησυχία. Σημείο 11. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ΚΑΜΑ. Έχουμε, όπως ξέρετε, συνάψει συμφωνίες με αρκετές χώρες ΑΚΕ. Βρισκόμαστε στο στάδιο της υπογραφής με αρκετές από αυτές και θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή μας, κύριο Λάμσταροφ, όμως σας παρακαλώ κάντε ησυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι και όσοι παραβίσκεστε στην αίθουσα, αγαπητοί συμμετέχοντες, θεατές, παρακαλώ μην ομιλείτε στην αίθουσα. Κύριε Λάμστορφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή με τις οικονομικές ε, συμφωνίες έχουμε φτάσει στο στάδιο που έχουν εξεταστεί όλες οι νομικές πτυχές. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ενοποίησης των κειμένων της συμφωνίας και αυτές οι συμφωνίες, όπως και οι άλλες, αφορούν τις οικονομικές μας σχέσεις με αυτές ε, τις ε, χώρες και την προσαρμογή τους στα πρότυπα του ΠΟΕ. Επίσης, αφορούν τη δημιουργία προοπτικών για αυτές τις χώρες, να βελτιώσουν τις εμπορικές τους ε, σχέσεις και συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 40 χρόνια είχαμε διμερείς σχέσεις με αυτές τις χώρες, οι οποίες βέβαια δεν οδήγησαν σε, ε, σε μεγάλη ανάπτυξη. Πολλές φορές μάλλον το αντίθετο. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, έχει μειωθεί, ε, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι συναλλαγέ μας λόγω του γεγονότος αυτού. Ε, αυτή η συμφωνία δεν είναι μόνο προ όφελο δικό μας, αλλά προ όφελο και των χωρών αυτών. Θα δώσει οικονομική ε, όθηση στις χώρες αυτές και θα βοηθήσει να εξαλειφθούν οι διάφορες ε, ασύμε, ασύμετρίες. και θα βοηθήσουν έτσι ώστε οι χώρες αυτές να ενταχθούν ομαλά στην παγκόσμια οικονομία. Οι ασυμμετρίες που έχουν παρατηρηθεί έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην αγορά, γι' αυτό οι συμφωνίες αυτές θα βελτιώσουν την ε, κατάσταση που αυτή τη στιγμή είναι εντελώς αντίθετη. Βρίσκονται αυτές οι χώρες σε μειονεκτική θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν ρήτρε ευελιξίας και επίσης υπάρχουν και διάφοροι μηχανισμοί εξασφάλισης ασφάλειας ε, των τροφίμων, διάφοροι μηχανισμοί που θα αφορούν τους βιομηχανικούς κλάδους και τα λοιπά σε αυτές τις συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, να τονίσουμε ότι σε αυτές τις συμφωνίες το πρώτο κεφάλαιο αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν σαφείς υποχρεώσεις για, όλους τους, ε, για όλα τα συμβαλώμενα μέρη να τηρήσουν τις ε, παγκόσμιες ε, συμβάσεις που θα προστατεύουν το περιβάλλον, θα προστατεύουν τα ε, εργατικά δικαιώματα. κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ε, ένα ψήφισμα με ε, έναν κατάλογο ο οποίος συμπεριλαμβάνεται εδώ στις συμφωνίες αυτές. Ε, πιστεύω πως ε, η η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρο ε, των επιθυμιών που είχε εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτό το ψήφισμα του 2009. τώρα, ένα πολύ σημαντικό πιστεύω όταν μιλάμε για τη διαδικαστία να δούμε ότι είμαστε σε ένα στάδιο που μπορούμε να καταφέρουμε πραγματικά αποτελέσματα. Η απόφαση για τις ε, υπογραφές πρέπει να ληφθεί από το Συμβούλιο. Αναμένεται να γίνει αυτό τον επόμενο μήνα, στην επόμενη σύνοδο. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία συνένεσης και αν καταφέρει το Συμβούλιο τον Ιούνιο να υπογράψει τη συμφωνία αυτή, τότε και εμείς θα έχουμε αρκετό καιρό, εμείς ε, όσο και οι άλλες χρόνες, για να κυρώσουμε τη συμφωνία πριν λήξει η ε, προθεσμία του Οκτωβρίου 2016, που είναι η προθεσμία που έχουμε τώρα. Αν καταφέρουμε δηλαδή πριν τον Οκτώβρη να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αυτή, τότε θα υπάρχει ένα καθεστώ πρόσβαση στην αγορά για όλε αυτέ τι χώρε. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε θα χωριστούν σε διάφορε ομάδε. GSP, MFA ή e EBA. Έχουμε διανύμει το χρονοδιάγραμμα στα μέλη της Επιτροπής. Στις 26 Απριλίου είχαμε μια πάρα πολύ ε, καλή συνάντηση με την ομάδα παρακολούθησης. Είχαμε ε, καλέσει εδώ τους ε, αρμόδιους διευθυντές που μας ε, παρουσίασαν τις σημαντικότερες πτυχές της συμφωνίας αυτής. Μετά είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα έχουμε μάλλον σήμερα τώρα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη συμφωνία και μετά τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε την έκθεση πριν τον Οκτώβριο δηλαδή. Αυτά λοιπόν ως προς τη διαδικασία. Με χαρά μου να ακούσω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους και όδης εισηγητές. Η κυρία Ραντς Καρσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο Γκάμπι Μάτο μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω σήμερα το πρωί, γιατί είναι κάπου αλλού σήμερα το πρωί και δεν μπορεί να παρεμπρεθεί και να σας πει ότι χαίρεται που προχωρούν ε, τα θέματα αυτής της συμφωνίας ε, και η συμφωνία συνάφηκε τις 15 Ιουλίου του 2014 με τις χώρες ΚΑΜΑ και έδωσε πέρα σε πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων. Ε, υποκαθιστά τη συμφωνία του 2009 που δεν ισχύει πια και είχαν υπογράψει το Λεσότο και η Μοζαμβίκη μεταξύ άλλων. Όπως λέει και ο κύριος Μάτα, η συμφωνία αυτή δίνει τέλος σε μια ε, περίοδο, μακρά περίοδο έλλειψης ασφάλειας δικαίου που ε, ήταν αντικείμενο ε, αμφισβήτησης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς ΠΟΕ για τη συμφωνία με τις χώρες αυτές. Όπως έλεγε ο συνάδελφος Λάμπστορφ, η συμφωνία προσφέρει πρόσβαση στην ασύμετρη αγορά για τις χώρες ΚΑΜΑ μπορούν να ε, προστατεύσουν από την ε, φιλελευθερωποίηση κάποιους ευαίσθητους ε, τομείς, να έχουν ρήτρες προστασίας, να προστατεύσουν αναδυόμενους τομείς. Υπάρχουν θέματα γεωγραφικών ενδείξεων που διευκολύνουν τις εξαγωγές και μπορούμε να έχουμε και ενίσχυση για την εξαγωγή στο εμπόριο μεταξύ των μερών και επίσης υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν δικαιώματα εξαγωγής για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε νέες επιχειρήσεις. Ε, και αυτά δείχνουν ότι υπάρχει σαφή συμμετρία με τη συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε ο εισηγητής. Η Μποτσουάνα, το Λεσότο, η Μοζαμβίκη, η Ναμίμπια θα έχουν πρόσβαση αφορολόγητα ε, για τις ε, μη δασμολογικούς φραγμούς, με εξαίρεση το εμπόριο όπλων φυσικά και επίσης ε, βελτιώνεται το εμπόριο με τη, σε σχέση με όσα εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει νέα πρόσβαση στην Τελωνιακή Ένωση της ε, Νότιας Αφρικής και θα έχει και μια συμφωνία με τη Μοζαμβίκη. Υπάρχει και μια ρήτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που δείχνει πόσο μεγάλη προσοχή προσδίζουν οι δύο πλευρέ ε, στα θέματα αυτά. Υπάρχει σχέση με τη Συμφωνία του Κοτονού, επομένω μπορούμε να κάνουμε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόσουμε και του κανόνε του Κοτονού. Και τέλο, ο κύριο Μάτο μου ζητά να επισημάνουμε την περιφερειακή διάσταση αυτή τη συμφωνία, η οποία συνάδει και με την Τελωνιακή Ένωση τη περιοχή, η οποία δεν παρακολύεται από αυτή τη συμφωνία. Θα είναι μια επιπλέον συμφωνία που θα προσθέσει κάτι παραπάνω σε αυτή την ένωση. Πρόκειται για κάτι το οποίο χαροποιεί ιδιαίτερα τον κύριο Μάτο, ο οποίο ε, ε, θέλει να σα το πω γιατί είναι από τα Κανάρια νησιά, μια εξόχω απομακρυσμένη περιοχή και ε, κυρίω τον ενδιαφέρει το θέμα των ζαχαροκάλαμων και η επεξεργασία σε ζάχαρη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ευρωπαϊκός κλάδος ε, των, της επεξεργασίας ζάχαρης με το τέλος των ποσοστώσεων και των εκχωρήσεων που έχουν δώσει σε, δοθεί σε άλλες χώρες ε, κινδυνεύει να εξαφανιστεί με ε, καταστροφικές συνέπειες για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Επομένως θεωρεί ότι είναι πονίδιστο ότι όλες οι συμφωνίες δεν ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Χαίρεται που αναφέρεται αυτό το μοντέλο σε αυτή τη συμφωνία και χαίρεται που υπάρχει συνέπεια στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ελπίζουμε να το υπάρχει αυτό και σε όλες τις ε, συμφωνίε. Και τέλος ο κύριος Μάτο χαίρεται για την τελική υπογραφή με όλες τις χώρες της περιοχής και την Νότια Αφρική, η οποία ε, δεν συμμετείχε στην ενδιάμεση εταιρική ε, συμφωνία. Μπορείτε να υποστηρίξετε λοιπόν, να βασίζετε συγγνώμη στην υποστήριξη του ΕΛΚ για τη συμφωνία αυτή. Ο κύριο Σούστερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όταν εξετάζουμε το θέμα αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι συμφωνίες οικονομικής ε, εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, ε, τις αφρικές κυβερνήσεις και κυρίως ε, τις χώρες της Νοτιού Αφρικής ήταν ακαθόδες ζήτημα για πάρα πολύ καιρό και αποσχολούσαν την κοινή γνώμη και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Ο λόγος γι' αυτό, και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε, είναι ότι ένα πολύ ε, φιλελευθερωποιημένο οικονομικό περιβάλλον ε, σε μία άνηση κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό είναι αυτό που ανησυχεί τους περισσότερους, γι' αυτό και υπάρχουν και αρκετές επικρίσεις και πρέπει να το έχουμε κατά νου στο παρελθόν πάντα διαπιστώναμε ότι υπήρχαν ε, πολλά μέτρα προστατευτισμού, ε, ρήτρε προστασίες και ε, πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη όμως προστασία. Ο κύριος Λάμστορ το επισήμανε αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο δεν εξετάζει το ελεύθερο εμπόριο, εξετάζει τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν η συμφωνία αυτή απλώς ως εμπορική συμφωνία. Πρόκειται για μια εταιρική ε, συμφωνία σύμπραξη ε, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι και σαφώς ε, γραμμένη στο κείμενο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να συνδεθεί και με άλλες πολιτικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό και τις μεταναστευτικές ροές, ε, τις οποίες αν θέλουμε να τις επιβραδύνουμε ή να τις σταματήσουμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αυτών των χωρών της Αφρικής. Και εγώ υποστηρίζω σαφέστατα αυτή την προσέγγιση. Πρόκειται λοιπόν για ισχυρισμούς και προκλήσεις ε, που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι να εξετάζουμε το θέμα της ε, βιωσιμότητας ε, πάντα. Δεν εξετάζουμε μόνο τα οικονομικά ζητήματα και να υπογράφουμε συμφωνίες. Πρέπει οι συμφωνίες αυτές να εφαρμόζονται καταλήλων, ως ε, να τις παρακολουθούμε και να τις αξιολογούμε και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και τη σχέση με τη Συμφωνία του Κοτονού. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερη σαφήνεια για πώς προτίθεται να γίνει αυτός ο έλεγχος και η παρακολούθηση. Επίσης πώς θα δημιουργηθούν οι δομές και στην κοινωνία των πολιτών αλλά και στις χώρες της ε, Νότιας Αφρικής. Και πώς θα διασφαλίσουμε δηλαδή ότι τα πιθανά λάθη θα μπορούν να διορθωθούν και να διαπιστωθούν από αυτούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης. Αυτά λοιπόν είναι τα απαραίτητα για μας, είναι τα σημεία στα οποία επίσης χρειάζονται διευκρινήσεις και αυτό που θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτές οι συμφωνίες για πολλές αφρικανικές χώρες ήταν κάτι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο. Και μάλιστα ορισμένες χώρες έχουν αντιρρήσεις, δεν θέλουν να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω πως μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και για τους μεν και για τους δε αυτή η ε, κύρωση να γίνει ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μην ε, έχουμε ενδεχόμενο να αρνηθούν σημαντικοί εταίροι μας στην Νότια Αφρική τη συμφωνία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν, ε, συνοψίζοντας, η συμφωνία μας δίνει πολλές ευκαιρίες, ταυτόχρονα όμως ε, περιέχει και αρκετούς κινδύνους, γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Έμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η συμφωνία αυτή, την οποία διαπραγματευθήκαμε με την ε, με τις χώρες ΚΑΜΑ χαροποιεί το ECR και περιμένουμε στην εφαρμογή της. Θα έχει πάει μεγαλύτερη ολοκλήρωση η Ευρωπαϊκή Ένωση με την περιοχή και καλύτερη συνεργασία κυρίως με τις χώρες αυτές. Αλλά πρέπει οι συμφωνίες αυτές να έχουν και ε, σαφή βάση στον ΠΟΕ θα μπορέσουν οι χώρες αυτές να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες ρήτρες ασφαλείας για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένους όγκους εισαγωγών ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες εισρωές που θα απειλήσουν κάποιους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε που υπάρχει και ένα αναλυτικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις τομείς του εμπορίου που θα την χάνουν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία δυνατοτήτων. Έτσι να μπορέσουν να οι χώρες αυτές από τις, ε, προτιμησιακό καθεστώ που του προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Χέλμουντ Σόλτ, για την ΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Μπέντ. Η ΚΟΥ έχει ακόμα πολλές ερωτήσεις για αυτήν την ε, συμφωνία. Από τη μία θεωρούμε ε, καλό το ότι μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στο πρώτο κεφάλαιο την βιωσιμότητα. Από την άλλη όμως δημιουργούνται πολλά ερωτήματα τα οποία θέλουν συζήτηση, ε, τα οποία αφορούν και άλλες συμφωνίες. Τι ε, γίνεται για παράδειγμα αν δεν ανανεωθεί η συμφωνία του Κοτονού. Θα μείνουμε στον αέρα, θα μείνουμε μετέωροι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γεφυρώσουμε το χάσμα. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία συνδέονται. Τι θα κάνουμε δηλαδή σε περίπτωση που δεν συνεχιστεί η Συμφωνία Κοτονού. Θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι πολλά από τα συμβαλώμενα μέρη σε αυτήν την συμφωνία είναι ικανοποιημένα με την ε, συμφωνία αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαφορές και αυτό ίσως οφείλεται στη διαφορά των δυνατοτήτων. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και πρέπει να αναπτύξουμε ένα τρόπο αντιμετώπισης. Πώς μπορούμε δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη να γίνει σε βάθος χρόνου και να διατηρηθεί. Είναι μια πολύ βασική ερώτηση για που αφορά πάρα πολλές χώρες της ε, Νότιας Αφρικής οι οποίες έχουν να επωφεληθούν άμεσα από μια τέτοια συμφωνία. Πρέπει όμως να απαντηθούν και ε, τα ερωτήματα έτσι ώστε η έκβαση πολιτική και οικονομική να είναι θετική ιδιαίτερα για τους πολίτες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι συμφωνίες έγιναν μετά από πίεση διαπραγματευτική 10 ετών και οι εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν δεν είναι σαφείς. Επίσης πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιο ρόλο παίζουν οι ελίτ αυτών των χωρών για αυτή την συμφωνία και πώς, μπορούμε να προετοιμάσουμε, πώς μπορούν να προετοιμαστούν μάλλον οι πολίτες για τις αλλαγές που θα ε, προκύψουν. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Γιούντιθ. Ε, πρόεδρε, ε, έχω πρόβλημα με, αυτό, με αυτή την ε, γνωμοδότηση, γιατί είμαι αντιπρόεδρος στην αντιπροσωπή, ήμουνα μάλλον στην προηγούμενη θητεία αντιπρόσωπο στην, αντιπροσωπή στην αντιπροσωπεία και μιλούσαμε για τους καλλιεργητές ζαχαροκάλαμου που ήθελαν την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές και είναι αδασμολόγητη η πρόσβαση στην αγορά. Αυτό είναι σημαντικό, συμφωνώ. Όμως από την άλλη, απαγορεύουμε τους ε, φόρους, εξαγωγικούς φόρους. Ενώ είναι εργαλείο αυτό του ΠΟΕ, περιορίζεται το πεδίο δράση ε, των ε, αναπτυσσομένων χωρών. Δεν έχουν κονδύλια. Επίσης, για αυτή την συμφωνία Ποιε επιπτώσει έχουμε για αυτέ τι συγκεκριμένε χώρε ενώ υπάρχουν και άλλε στα πλαίσια περιφερειακή συνεργασία με διαφορετικέ χώρε τη ΚΑΜΑ, ε, όπου οι επιπτώσει είναι πολύ διαφορετικέ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ διαφορετικέ οι οικονομικέ συνθήκε και το επίπεδο οικονομική ανάπτυξη ανάμεσα σε αυτέ τι χώρε. Ε, η, Νότια Αφρική έχει μέσα εισόδημα. αυτέ οι χώρε είναι λιγότερο ανεπτυγμένε είναι λάχο, οπότε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τι ίδιε συμφωνίε. Ε, τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις χώρες. Εγώ προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί τους. Ε, δεν έχω περι... παραπεριορισμένες πληροφορίες ε, και συνεχίζω να ψάχνω. Και τέλος, πριν από λίγες εβδομάδες η Επιτροπή μας συζήτησε εδώ μια μελέτη για τις επιπτώσεις ε, το, τη συμφωνίες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συγκεκριμένα για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών ε, και προκύπτει ότι διευκολύνεται το ξέπλυμα χρήματος μέσα από αυτές τις συμφωνίες ε, και μην ξεχνάμε το ρόλο αυτών των χωρών και όταν γίνονται έρευνες για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ε, η Νότια Αφρική είναι δέκατη στη σειρά σε σχέση με τις εξαγωγές ε, νομιμοποιημένων παρανόμων εσόδων. Ποια, ποια λοιπόν η επίπτωση μια τέτοιας ε, συμφωνίας, εάν η νομιμοποίηση εσόδων έχει μια νέα, ένα νέο πεδίο δράσης, αν θέλετε, δηλαδή μια νέα αγορά, τη βρίσκω ένα ανησυχητικό το περιεχόμενο της συμφωνίας. Δηλαδή, για να αποφασίσω, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ, Τζουντ. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει, που εξετάζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. Ε, δεν θα πρέπει να νιώθουμε ότι τελούμε υποπίεση για την πρόσβαση στην αγορά, για τον κανονισμό αυτό. Δεν ε, πήγε, δεν χρειάζεται να λάβουμε ε, ταχύτατα την απόφαση, οπότε να μην αφήσουμε να μας ασκήσουν πίεση. Και επειδή είναι τόσο σημαντική αυτή η απόφαση, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μόνο τη διαδικασία στην απόφαση, αλλά να συνοδεύσουμε την απόφαση με την έκθεση, γιατί είναι έγκυρα αυτά τα σχόλια που ακούμε από τους συναδέλφους και θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την γνωμοδότηση για την βιώσιμη ανάπτυξη και Αυτό είναι το, ε, το μη το αν θέλετε, ε, αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία σε σχέση με τι άλλε που θα τεθούν ενισχύ. Όμω είναι περιορισμένα τα θετικά αποτελέσματα και αυτέ οι έξι χώρε έχουν επικυρήσει τις 8 ε, βασικές συμβάσεις σε Διεθνούς ε, ε, Γραφείου Εργασίας. Το βασικό όμως είναι πώς εφαρμόζονται στην πράξη, γιατί δεν υπάρχουν δομές παρακολούθησης. Τα είπε και η Τζόντι. Δεν έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας για να φροντίσουμε να γίνει σωστά η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν λάβει σχέση με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, Κορέα, Κολομβία, Περού. Οι αντίστοιχε συμφωνίες έχουν πολύ ψηλότερες προδιαγραφές και μία συγκεκριμένη χώρα με απασχολεί ιδιαίτερα διότι το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί για τη Σουαζιλάνδη συγκεκριμένα. Εγκρίναμε γνωμοδότηση στην Ολομήλη πριν από ένα χρόνο, όπως θα θυμάστε και ξεκάθαρα. Είπαμε πως οι φυλάκες των πολιτικών ακτιβιστών και η κατάργηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων συνιστά κατάφορη παραβίαση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Σουαζιλάνδη βάζει του κεφαλαίου βιώσιμη ανάπτυξη σε τι συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση ε, χωρών ΚΑΜΑ ε, και η υποστήριξη του Κοινοβουλίου θα είναι συνάρτηση τη στήριξη αυτών των υποχρεώσεων ε, που έχει αναλάβει ο Ζελιλάδη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε πρώτο. Ζητήσαμε επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένε προτάσει για την παρακολούθηση. Ε, πολύ ωραία, εύσχημα λόγια. Τίποτα όμω γραπτό, τίποτα συγκεκριμένο καμία πρόταση και νομίζω ότι αυτή την πρόοδο θα πρέπει να διαπιστώσουμε η δύο ισόμωση προτού εγκρίνουμε ή απορρίψουμε αυτή την έκθεση. Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ. Ε, έχω ακόμη ερωτηματικά για αυτές τις ε, συμφωνίες. Ε, πρώτον, ακούμε συχνά την επιχειρηματολογία θα πρέπει να τηρήσουμε τις προδιαγραφές του ΠΟΕ. Το είπε η Τζοντή, δεν υπάρχει καμία καταληκτική ημερομηνία και στα πλαίσια του γύρου της, της Ντόχα στον ΠΟΕ, ούτως ή άλλως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είχαν καταθέσει παρατηρήσεις για αυτές τις συμφωνίες και τελικά όμως δεν ελήφθη τίποτα υπόψη για αυτές τις χώρες. Εμείς τι θέλουμε, όχι να αντικρούσουμε τις διεκδικήσεις αυτών των ε, χωρών, αλλά να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν. Και δεύτερον, αυτή η ασύμμετρη ανάπτυξη αληθεύει πως η συμφωνία με τις χώρες ΚΑΜΑ ε, όντως ε, βασίζονται σε αυτή την ασύμετρη ε, απελευθέρωση. Όμως υπάρχουν προϊόντα που αποκλείονται από αυτές τις συμφωνίες. Και τι διαπιστώνουμε, ότι με διαφορετικό τρόπο μπαίνουμε σε αυτή την περιοχή. γιατί την Νότια Αφρική, ε, Βόρειο κρέας, την μπανάνες, παραδείγματο χάρη, αλλά το επιτρέπουμε για την Μποτσουάνα. Δηλαδή ανοίγουμε πόρτες και παραθυράκια σε διαφορετικές χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι να ε, καθιερωθούν ε, περιφερειακές διαφορές και μην ξεχνάμε ότι είναι 16 χώρες χώρες συνολικά και αυτή η συμφωνία λοιπόν ε, αφορά μόνο 6 χώρες. Άλλη οργάνωση περιφερειακή έχουν αυτές οι χώρες από πλευρά τους και άλλοι προσπαθούμε να επιβάλλουμε εμείς. Ε, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η Τζούντιθ, ούτε ο Ιωακήμ, αλλά μιλάμε και για τις διαφορές με τη Συμφωνία Κοτονού που εκπνέει το 20 θα υπάρξει περίοδο μετά το Κοτονού, Όμω το 2016 αναφερόμαστε στην ε, Συμφωνία Κοτονού που εκπνέει σε τέσσερα χρόνια. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα εκπνεύσει και δεν υπάρχουν μέσα από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόσθετα κονδύλια για να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε. Επίση, ε, το 2009 παραπέμπουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν έχω πρόβλημα και 25 χρόνια πίσω να είναι γνωμοδότηση, κανένα πρόβλημα. Το 2016 όμω μήπω θα έπρεπε να προσαρμόσουμε την πολιτική στάση του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτέ τι συμφωνίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντεσαρνές, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρ Λάμστροφ, διότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη έκθεση και θα πρέπει να ε, εξαντλήσει την ευφυΐα και την ε, ε, διακριτικότητά του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Λοιπόν, θα σταθώ σε κάποια θέματα στα οποία αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι. Πώ μπορούμε καταρχά να κάνουμε του Αφρικανού να νιώσουν ότι δεν του επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία. Γιατί αυτή την αίσθηση έχουν αυτή τη στιγμή, ότι εδώ και χρόνια του επιβάλλουμε πράγματα. Ενώ πρέπει να νιώσουν ότι αυτή η συμφωνία είναι δική του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Θα πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι προ το συμφέρον του και να επενδύσουν στο περιεχόμενο αυτή της συμφωνίας για να πούνε να εμείς αυτό θέλουμε ως Αφρικανοί και για τις χώρες μας αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, θεωρώ ότι επαφείται σε εμά ως Ευρωπαίους να ε, δούμε ότι η ανοικοδόμηση της Αφρικής δεν είναι θέμα εμπορίου ή μείωση των δασμολογικών φραγμών. Ε, πρέπει να υπάρχει αυτάρκεια, για παράδειγμα, για τη γεωργία σε κάποιε Αφρικανικέ χώρε, οι οποίε πρέπει να έχουν μια γεωργία και όχι να ε, ε, δημιουργούν την απόλυτη ένδυα στις ε, μεγάλες αφρικανικές πόλεις λόγω εξάντλησης των ποσοστώσεων που έχουν. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα βιομηχανικό κλάδο, θέματα ενέργειας, περιφερειακή ολοκλήρωση, απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Πρέπει λοιπόν από αυτή την άποψη να δούμε το θέμα γιατί έχουμε Ευρωπαίους και Αφρικανούς, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα με μια λίγο διαφορετική λογική. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Σάντρα, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε που συμπεριλάβατε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο με καλέσατε. Καταρχάς ε, να σας πω ότι εάν δεν παραταθεί η Συμφωνία Κοτονού, κύριε Σόλτς, οι βασικές αρχές είναι ε, εγγεγραμμένες στην Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Δηλαδή, η διαδικασία του Κοτονού μπορεί να εκπέσει, αλλά μπορεί να επιβάλλει κυρώσει για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διότι αναφέρονται σε αυτή τη συνθήκη. Και εγώ θα προτιμούσα να υπήρχαν και τα δύο προσωπικώς. Αυτή βέβαια δεν είναι επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εν τέλει τι δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε τις διαδικασίες. Στο Κοτονού υπάρχει η διαδικασία των 90 ημερών, υπάρχει το άρθρο 96, εδώ θα επιβάλλουμε κυρώσεις μονομερούς. Τουλάχιστον να είναι σαφές ε, τι θα χάσουμε. Για τους ε, το, φόρους εξαγωγές, κυρία Αρχεντίνη, σας ε, παρακολουθούσα πολύ προσεκτικά, γιατί νομίζω ότι μιλάτε από καρδιάς και όντως αυτές οι ε, Εταιρική σύμπραξη ε, μας αφορούν όλους. Ε, αρχίζουν να λήγουν σιγά σιγά αυτοί οι φόροι εξαγωγές γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και νόμοι που ε, ε, θεμελιώνονται στην, στους φόρους εξαγωγής στις χώρες αυτές. Μπορεί εμείς να μην διαβημάζουμε κατάλληλα το μήνυμα αλλά οι Αφρικανοί έχουν αντιληφθεί ότι έχει αλλάξει η συμφωνία στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Περιφερειακή συνεργασία. Έχετε δίκιο. Γιατί η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ είναι διαφορετικά πράγματα οι χώρες ΚΑΜΑ, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι χώρες αυτές έχουν επιλέξει τις περιφέρειές τους. Όλες αυτές οι συμφωνίες τη οικονομικής εταιρική σχέσης έχουν συμφωνηθεί από τις ε, ίδιες τις χώρες. Και έχουμε ξεκινήσει ήδη τι συζητήσει. Ε, και ε, στρατηγικές εθνικής εφαρμογής της ε, Συμφωνίας Εταιρικής σχέση Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να χτίσουμε γέφυρες και σε αντίθεση με αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί χαίρομαι που έχω συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ που έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις. Επίσης, ε, όπως είπατε κι εσείς, ε, ε, υπάρχει το πρόβλημα της Μοζαμβίκης. Αλλά η Μοζαμβίκη έχει τελείως διαφορετική προσφορά, προσφέρει πολύ λιγότερα, προσφέρει 74% και επομένως διαφέρει από τις υπόλοιπε χώρες. Νομοποίηση παρανόμων εσόδων. Πολύ καλή παρατήρηση. Όντω είναι πολύ μικρέ αυτέ τι συμφωνίε ακόμα, αλλά χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα και νομίζω ότι και οι ίδιε οι χώρε θα ε, προσπαθήσουν να επεκτείνουν κι άλλο τις συζητήσεις βάσει της συμφωνίας. Εμπιστεύομαι τους εταίρους μας ότι πραγματικά θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Μπορεί να μην είναι μεγάλο εργαλείο όσον αφορά την ε, ισότιμη κατανομή του πλοίου του και εδώ να έρθω σε αυτό που λέει ο κύριος Σούστορ, σίγουρα είναι άνηση αυτή η κοινωνία. Ε, δεν υπάρχουν ε, οικονομικά από την κορυφή προς τη βάση και ίσως ε, να θεωρήσουν οι ίδιες οι χώρες ότι αυτές οι συμφωνίες μπορούν να τους βοηθήσουν. Σίγουρα δεν θα είναι πανάκια για τα πάντα. Ως προς το γεγονός ότι δεν υπάρχει πίεση τρόπον την εγώ θα έλεγα ότι εξαρτάται από το πρίσμα. Αυτές οι χώρες ε, έχουν διαπραγματευτεί πολύ προηγμένες συμφωνίες υπέρ της ανάπτυξης που έχουν πάρα πολλά ωφέλη για αυτές. Εάν λοιπόν δεν δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους, δεν θα μπορέσουν για παράδειγμα να επωφεληθούν από τους νέους κανόνες γεωγραφικών ενδείξεων που υπάρχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις περιφέρειες. Το να τα συσσωρεύσουμε όλα μαζί είναι κάτι διαφορετικό βεβαίω. Και επίσης θεωρώ ότι θα θεωρήσουν ότι είναι πάρα πολύ κακό σημάδι αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα επανέλθω σε αυτό. Διότι ε, μας βλέπουν ως ε, ε, αυτούς που τους υποδέχονται εδώ. Μπορεί βέβαια να μην τα έχουμε καταφέρει ακόμα με τη Σουαζιλάνδη, έχετε δίκιο, αλλά χάρη στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση, χάρη στη μόχλευση που υπάρχει και χάρη στι εξαιρετικέ συνεδριάσει και τα όσα έκανε η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ με του υπουργού από τη Σουαζιλάνδη, έχει αρχίσει να υπάρχει κάποια κίνηση από πλευρά του. Μπορεί να μην τα έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά βλέπω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή και για του ε, τα όσα είπε ο πρόεδρος Λάγκε στην αρχή, για την εξωτερική πολιτική δηλαδή, όχι μόνο για το εμπόριο και σε αυτές τις συμφωνίες. Τώρα, μια διαφορετική είσοδο, δηλαδή αγαθά τα οποία μπαίνουν σε μια χώρα και πηγαίνουν σε άλλη. Αυτό τελικά θα ήταν απάτη. Ε, εγώ έχω εμπειρία σε αυτό και δεν είναι κάτι δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε και το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Το γεγονό ότι επιβάλλουμε συμφωνία στου Αφρικανού, κυρία Ντεσαρνέσε, ναι, αυτό ήταν αυτό το οποίο πρεσβεύαμε στο παρελθόν. Ε, Εχθέ συζητούσαμε και τον υπεριαλισμό με κάποιον ε, συνάδελφό σα, ο οποίο είχε μια συνάντηση μαζί μα και πρέπει να σα πω ότι έχει αλλάξει η αφήγηση. Εμεί ε, δεν του το έχουμε επιβάλει, είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε αυτέ συμφωνίες. Υπάρχει βέβαια η κοινωνία των πολιτών που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά επιτρέψτε με να πω ότι αυτό το οποίο βρήκα το 2009 πόρο απέχει από αυτό το οποίο ισχύει σήμερα. Και επίση να σας πω ότι ε, δίνοντας τη σύμφωνη γνώμη μας ε, και ε, καλωσορίζοντας αυτούς τους ανθρώπους τώρα, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι προσπαθούμε να του εκμεταλλευτούμε. Ε, αν προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση για να προωθήσουμε κάτι καλό, θα ήταν ό,τι καλύτερο για αυτέ τι χώρε. Πραγματικά λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να του δώσετε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα Συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Τηρήσατε και το χρόνο. Καταπληκτικά. Ο κύριο Λάμστροφ. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτέ τι πρώτε αντιδράσει. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία γιατί οι λεπτομέρειες αυτές ε, συζητήθηκαν. Σωστά είπε ο κύριος Σούστερ ότι η κοινωνία των πολιτών έχει μεγάλο ενδιαφέρον και την έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό. Ε, η κυρία Ντάρλινγκ είπε ότι το κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα είναι το καλύτερο ή τουλάχιστον το λιγότερο κακό ε, σε αυτή τη συμφωνία. πρέπει να δούμε τι μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή τη συμφωνία από τη δική μας πολιτική ατζέντα. Τι μπορούμε να επιτύχουμε με μια τέτοια συμφωνία. Και εδώ αξίζει να προβληματιστούμε για το αν ζητάμε πάρα πολλά, αν θα φορτώσουμε τη συμφωνία με ε, πολλά πράγματα τα οποία στο τέλος θα οδηγήσουν σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Είναι αυτό που είπε και η κυρία Ντεσσαρνές. Κανείς δεν πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή από μόνη της θα είναι επαρκής έτσι ώστε να δημιουργήσει, να χαράξει νέα, ε, νέους δρόμους για ανάπτυξη. Μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό στην καλύτερη περίπτωση, όμως ε, η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει και ε, σωστές ε, βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων, των οικονομικών συνθήκων και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μία μόνο συμφωνία. Μετά η κυρία Αρένα αναφέρθηκε στο ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων σε αυτές ε, τις ε, χώρες και ότι δεν μπορούμε να ε, έχουμε μία συμφωνία για όλα και επίσης ότι οι χώρες αυτές έχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Αυτό πιστεύω πως δεν είναι κάτι που είναι επικριτικό προς τη συμφωνία αυτή, αλλά πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σωστό. Επίσης, η συνάδελφος από το ΕΛΚ μας είπε ο, για το τέλος της αβεβαιότητας που έχει έρθει. Εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου μέσω της συμφωνίας αυτής σε αυτές τις χώρες ή να βελτιωθεί τουλάχιστον η κατάσταση. Όπως είπε η Μαρίνα Αρένα, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν αποχωρήσει, που έχουν ένα opt-out. Η Αγγόλα, ας πούμε, δεν έχει υπογράψει. σε αντίθεση με άλλες ε, χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε επίσης όρις και να σεβόμαστε τους ε, εταίρους μας στην Αφρική. και να μην τους ε, υποτιμούμε, να μην τους εκβιάσουμε να υπογράψουν. Μετά, ε, διατυπώθηκε το ερώτημα του τι γίνεται με το μηχανισμό παρακολούθησης. Ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Και καταρχάς υπάρχουν μηχανισμοί στα πλαίσια της συμφωνίας, υπάρχει ένα συμβούλιο, υπάρχει μια ομάδα διοικητικών η οποία θα ασχολείται ακριβώς με αυτό, υπάρχει η συμφωνία του Κοτονού που δημιουργεί ένα πλαίσιο όμως σίγουρα υπάρχει χώρος και περιθώριο για βελτίωση και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε διότι όντως είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικά κείμενο, μια σημαντική συμφωνία και αν θέλουμε να επιτύχουμε πραγματικές ουσιαστικές βελτιώσεις πρέπει να το ε, εφαρμόσουμε. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αναμένω με αγωνία τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμστορφ. Πρέπει να δημιουργηθεί σίγουρα το σωστό φόρουμ συζήτησης για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτούς τους ε, μηχανισμούς. Τις 15-16 Ιουνίου θα συζητήσουμε την συνέχεια της έκθεσης αυτής για να δούμε και πώς θα προχωρήσουμε. Και μετά τις θερινές διακοπές ε, θα πάμε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 18. Έχουμε μια δημόσια ακρόαση για το Διεθνές Ψηφιακό Εμπόριο, η οποία θα αρχίσει τώρα με μια μικρή καθυστέρηση, ωστόσο όμως με μεγάλη αποφασιστικότητα και ενέργεια. Εάν κάποιος θέλει παραδόξω να εγκαταλείψει την αίθουσα, κάτι που δεν θα καταλάβω, διότι η ακρόαση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, τότε σας παρακαλώ να το κάνετε με ησυχία. Ησυχία. Το ψηφιακό εμπόριο είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και εξελίσσεται ταχύτατα. Έχει τεράστιο δυναμικό για ανάπτυξη και απασχόληση. Είναι όμως και ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, διότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι πρέπει να διέπουν το ψηφιακό εμπόριο. Και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Δεν θα κάνω κανένα άλλο εισαγωγικό σχόλιο, αλλά θα καλέσω αμέσως τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε δύο πάνελ σε αυτή την ακρόαση. Το πρώτο αναφέρεται στο δυναμικό και το δεύτερο στους κανόνες. Και στα δύο πάνελ έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες. Το πρώτο πάνελ θα έχει καλέσει με τον Ρόμπερτ Σλέγκερμιλχ ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει έρθει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και τον Τζόσουα Μέλτσερ από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins Εδώ είστε. Καλημέρα. Για να συζητήσουμε λοιπόν το δυναμικό του ψηφιακού εμπορίου. Θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Σλέγγελμιλχ για 10 λεπτά. Στη συνέχεια στον κύριο Μέλτσερ και μετά στους συναδέλφους, τα μέλη της Επιτροπής, ο καθένας για ένα λεπτό για ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σε αυτά τα 10 λεπτά να σχολιάσω το ζήτημα από τη σκοπιά της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εμπορίου, να μιλήσω για το τις προοπτικές, αλλά νομίζω οι συνάδελφοι έχουν πολύ περισσότερα, ε, πολλά περισσότερα στοιχεία σε σχέση με αυτά που κάνουμε και θα ήθελα επίσης ε, να μιλήσω για την προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε σε αυτό το εξόχως σημαντικό ζήτημα. Όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε ε, με ποιο τρόπο η ψηφιακή επανάσταση καταρρύπτει τα γεωγραφικά εμπόδια, τα, την απόσταση που μας χώριζε και στη γάμα δέλτα ε, εμπορίου αλλάζουν, όπως διαπιστώνουμε, και τα ε, όσα γνωρίζαμε για το εμπόριο στο παρελθόν. Δημιουργούνται όμως ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες, κυρίως για μικρές επιχειρήσεις. Ε, λύνονται κάποια από τα προβλήματά τους ε, για τα ταξίδια στο χώρο και στο χρόνο. Να δώσω και κάποια στοιχεία. Ε, το συνολικό εμπόριο, που μεταβίαση υπήρχε πριν από 25 χρόνια, ανέρχεται σε 12-3 ευρώ πλέον. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα στοιχεία για την ψηφιακή οικονομία βλέπουμε για την περίοδο 2010 έως 2016 όπου ε, σημειώθηκε η κρίση σχεδόν σε όλους τους τομείς, ε, αναμένεται ότι θα φτάσουμε στο 5,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για το 2016 ε, κατά διαστολή με το 3,8% το 2010. Βλέπετε σε πραγματικούς όρους πόσο ε, σημαντική αλλαγή, ριζική αλλαγή σημειώνεται σε αυτό τον ε, τομέα. Υπάρχουν ανησυχίες για την υπεροχή ε, στη νέα τάξη πραγμάτων, να το πω έτσι, των αμερικανικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι στην Ευρώπη έχουμε σχετικά καλές επιδόσεις. Δηλαδή, στο σύνολό της η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ε, των ψηφιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών δηλαδή που προσφέρονται ε, ψηφιακά και που ποσοτικοποιούμε. Σχεδόν το 1 τέταρτο των εξαγωγών μας είναι υπηρεσίες 465 δις δολάρια και τα λέω σε δολάρια γιατί οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτά τα στοιχεία ε, βάσει των μελετών ε, και 390 ε, δις αντίστοιχα για το ΣΥΠΑ. Βέβαια τα στοιχεία είναι από το 12. Είναι μεγάλο το δυναμικό στην Ευρώπη τα καταφέρνουμε σχετικά καλά. Το θέμα όμως είναι γιατί πράγμα μιλάμε τελικά ε, με αυτές τις ε, λέξεις ε, ψηφιακό εμπόριο. Λοιπόν, για μας, στη δική μας Γενική Διεύθυνση, Νομίζω ότι πρέπει να ε, το χωρίσουμε σε διαφορετικά τμήματα που μπορούμε να διαχειριστούμε. Δηλαδή, ε, να έχουμε μικρά τμήματα τη ψηφιακή οικονομία, τα οποία πιο εύκολα θα διαχειριστούμε και έτσι να αποκομίσουμε τα οικονομικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμω να διαφυλάξουμε και του βασικού κανόνε λειτουργία μα. Θα προσπαθήσω λοιπόν μέσα από παραδείγματα να καταδείξω ακριβώ ε, αυτή την ανάγκη. Πρώτον, το πλέον αμφιλεγόμενο ζήτημα και δύσκολο είναι τα δεδομένα και οι ροέ δεδομένων. Το δυναμικό που έχουμε της χρήσης των δεδομένων είναι πελώριο, ε, ταυτόχρονα όμως ε, μας φέρνει αντιμέτωπους με δυσκολίες. Ας ε, μην ξεχνάμε όμως ότι αυτός είναι ο πυρήνας του εμπορίου, μετακίνηση δεδομένων και ορισμένες φορές μας το παρουσιάζουν ως ε, κάτι που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Όχι, για την Ευρώπη, για όλες τις χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν είναι πολύ σημαντικό. Πολύ απλά παραδείγματα θα σας δώσω για να το αποδείξω. όταν ε, σηκώνετε λεφτά στη ΣΥΠΑ ή οπουδήποτε αλλού, μεταφέρετε δεδομένα γιατί πρέπει να ταυτοποιηθεί η κάρτα σας, η πιστοτική. Επίση, οι στόλοι των φορτηγών, παραδείγματο χάρη, οι αισθητήρε ε, φέρνουν στοιχεία ακόμη και για την ε, συμπεριφορά του οδηγού ω ε, προς τη νομοθεσία για το περιβάλλον. Όλα αυτά πηγαίνουν στα κεντρικά και αναλύονται ω δεδομένα παραδοσιακές υπηρεσίε, ασφάλειες, όλα αυτά μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά. Και έχουμε και τα, τους κλασικούς τομείς ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή όταν αγοράζουμε επιγραμμικά, ε, αυξάνονται οι συναλλαγές ε, ως προς την εφοδιαστική, ως προς τους πελάτες, ε, μεταβιβάζονται συνεχώς δεδομένα. Τι γίνεται με την ανάλυση των δεδομένων. Όλες αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τι τις κάνουμε τελικά για τους πελάτες, για το μάρκετινγκ, για τη χρηματοδότηση, για τους ανθρώπινους πόρους, όλα αυτά συνυπολογίζονται και ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ροές γίνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό ε, μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια εικόνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και για την ηλεκτρονική υγεία. Μεγάλο ανεπενταλευτό, δυναμικό. Δεν χρειάζεται να είσαστε ε, γιατρός ε, για να έχετε καλή διάγνωση, παιδεία, επιγραμμική. Πολλές υπηρεσίες ψηφιοποιούνται και θα σταματήσω εδώ. Ήθελα μόνο να έχετε μια ιδέα για το τι πράγμα μιλάμε τελικά όταν το θέμα μας είναι το ψηφιακό εμπόριο και όλα αυτά συνδέονται άμεσα με την ροή των δεδομένων. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκαθάριζε στο ψήφισμα για την ΤΙΖΑ και για την ΤΙΤΙΠ ότι δεν θέλουν να υπονομευθούν τα πρότυπα για τα προσωπικά δεδομένα. Όμως όλα επιστρέφουν σε αυτό τον πυρήνα. Ε, θα πρέπει φυσικά να συμμορφωθούμε με μελλοντική νομοθεσία για την ιδιωτική ζωή, για τη μεταφορά των δεδομένων Ξέρετε όλοι ε, ε, τι ε, λέγεται για την προάσπιση της ιδιωτικής σφαίρας και στην ψηφιακή οικονομία. Δεν θα έχουμε ρήτρε που θα λένε ανάλογα με το τι συμφωνήσατε εσείς ή οι εταίροι σας για τα ιδιωτικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να έχουμε κανόνες για την μεταβίβαση δεδομένων. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ιεράρχηση των κανόνων. Ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επειδή ε, ε, ασχολούμαι πολύ καιρό με αυτό το ζήτημα θα δώσω ένα παράδειγμα. Από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προέρχονται όλες αυτές οι νομοθετικές διατάξεις και όλα αυτά χρονολογούνται από το 90, από τον ΠΟΕ. Τότε οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, από τότε ε, ήταν για τις τράπεζες ε, και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τότε υπήρχε ήδη το πρόβλημα με των προσωπικών δεδομένων και είχαμε λοιπόν το, τη συμφωνία για τις υπηρεσίες του ΠΟΕΜ και τα παραρτήματα και κάποιε συμφωνίε εμπορικέ με την Κορέα παραδείγματο χάρη. και έχουμε ήδη κανόνε για τη ροή δεδομένων και την προστασία ε, των ε, ατομικών δεδομένων και τη ιδιωτική σφαίρα. Ε, Τέλο πάντων, γιατί πέρα από τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, αυτό το φάσμα των νομοθετικών διατάξεων επισέρχονται σε όλους τους τομείς πλέον και αν δείτε την τελευταία ανακοίνωση που κάναμε τονίζουμε πόσο μεγάλη, πόσο μεγάλη προτεραιότητα είναι για εμάς ε, στο μέλλον να ρυθμίζουμε με τον πλέον ενδεδειγμένο, πλέον πρόσφορο τρόπο τις ε, μεταβιβάσεις, τις ροές δεδομένων. ακούμε πολλά για τη ροή ε, δεδομένων προς τη ΣΥΠΑ. Δεν είναι αυτό το βασικό μας πρόβλημα. Το ένα από τα μεγαλύτερα άλλα προβλήματά μας ε, είναι η ροή δεδομένων προς όλες τις υπόλοιπες χώρες. Πολλές χώρες σε διάφορες περιοχές του κόσμου ακολουθούν νομοθεσία που ε, ουσιαστικά ε, κρύβουν ένα προστατευτισμό και η προστασία των δεδομένων γιατί θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί των συναλλαγών και και επιβάλλουν να ε, προσδιορίζονται γεωγραφικά τα δεδομένα για λόγους που εμείς θεωρούμε ανάρμοστου. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί έτσι χάνουμε πολλές εμπορικές συναλλαγές. Δεν θα μπορούμε να συμμετάσχουμε ε, καν σε ψηφιακή οικονομία αν για τα μηχανήματα ή για τέτοια προϊόντα δεν εξασφαλίσουμε μια ανεμπόδιστη ε, ροή δεδομένων. Αυτό είναι ένα τμήμα του πρόβλημα αλλά έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Άλλο 1,5 λεπτό έχω και θα το χρησιμοποιήσω για να πω το ψηφιακό εμπόριο σημαίνει και άλλα ε, πράγματα, ε, υπηρεσίες ε, τηλεπικοινωνιών, γιατί είναι η τεχνολογία, ευρυζωνικές συνδέσεις με ε, ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού για την πρόσβαση ε, στις γραμμές. Ε, δεν μπορού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές λοιπόν που έχει ο, η, η εταιρεία διαχείρισης, τότε έχετε πραγματικό πρόβλημα γιατί δεν έχετε πρόσβαση στην υποδομή. και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, υπάρχει και το πρόβλημα της εμπιστοσύνης, γιατί έχουμε τους κανόνες για το spam, παραδείγματος χάρη, spam, anti-spam, τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών ε, όταν μπαίνω σε ένα κατάστημα ή το ίδιο όταν αγοράζω επιγραμμικά μπορώ να το επιστρέψω. Ποιες, ποιοι κανόνε ε, ισχύουν. Υπάρχει ένα τμήμα του κεκτημένου τη εσωτερική αγορά που δεν θα μα αποσχολήσει σήμερα, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι συνιστά πρόβλημα και για την ψηφιακή οικονομία, γιατί θα πρέπει να τα εξετάσουμε από την σκοπιά του ίντερνετ. Ε, και οι εξωτερικοί κανόνε θα πρέπει όχι μόνο να είναι συμβατοί, αλλά να ε, μα οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση που επιδιώκουμε. Και επίση για τις αγορές, για τις πωλήσει, ε, για την προστασία των προσωπικών ε, δεδομένων. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό τμήμα του ε, ηλεκτρονικού εμπορίου, ότι ισχύει για τους παρόχους υπηρεσιών πώς προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες η πλατφόρμα. Έληξε και ο χρόνος μου. Θα σταματήσω εδώ. Είναι πολύ μεγάλο το ε, ανεκμετάλλευτο δυναμικό και ε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ε, και βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από άλλες περιοχές του κόσμου σε σχέση με το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε την ψηφιακή οικονομία. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάλιστα από την Σχολή Τζον Χόπκινς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε εδώ ε, να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να σας ε, πω για τα ψηφιακά ζητήματα για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργούν τα ψηφιακά δεδομένα για το διεθνές εμπόριο και τις θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο προκειμένου να συμμετέχουν στην παγκόσμια οικονομία με τρόπους που δεν μπορούσαν στο παρελθόν. Επομένως, πρόκειται για μια συναρπαστική εξέλιξη. Θα προσπαθήσω στο δεκάλυπτο που μου δίνετε να σας πω κάποια πράγματα για το γιατί συμβαίνουν αυτά και τι γίνεται με τις ροές δεδομένων για τα οικονομικά και το εμπόριο και τις δυνατότητες που υπάρχουν ε, για τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγούνται του τομέα. Όπω είπε και ο συνάδελφο, οι ροέ δεδομένων ουσιαστικά διέπουν το πώ λειτουργεί η οικονομία, οι εφοδιαστικέ αλυσίδε, οι επιχειρησιακέ ε, συναλλαγέ ε, γίνονται χάρη στη δυνατότητα ανταλλαγή δεδομένων παγκοσμίων. Τα δεδομένα εξαρτώνται από το διαδίκτυο, αλλά δεν περιορίζονται μόνο αυτό, σε αυτό. Ε, ρέουν και στο λεγόμενο βιομηχανικό διαδίκτυο εντό των επιχειρήσεων. Μπορεί να είναι λογισμικό όταν ε, κατεβάζουμε λογισμικό, μουσική, βίντεο, αλλά διευκολύνει και το εμπόριο όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα για να έχουμε πρόσβαση στα ε, συσκευέ επικοινωνία μα ή στο ηλεκτρονικό μα ταχυδρομείο. Έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο ροές δεδομένων από, για το παγκόσμιο ΑΕΠ από το εμπόριο αγαθών. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο είναι καταρχάς από την αλλαγή των οικονομικών και επίση, το γεγονό ότι κάνουν πιο παραγωγικέ τι επιχειρήσει στις διεθνεί αγορέ, και όπω είπε και ο συνάδελφο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την οικονομία, όχι μόνο τον τομέα τη πληροφοριακή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσει σήμερα, είτε είναι στο μεταπληκτικό τομέα, στη γεωργία, στην έρευνα. Ε, οι σύγχρονε επιχειρήσει χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τι συναλλαγές του, για τις ε, ανταλλαγέ του και θα επηρεάσουν όλο ένα και περισσότερο το διεθνέ εμπόριο. Το ανταγωνιστικό πλέον ε, έκτημα είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιείται το βιομηχανικό ε, διαδίκτυο και θα χρησιμοποιείται και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέλλον. Επίσης δίνεται πρόσβαση σε πελατολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακό και έτσι οι πλατφόρμες του διαδικτύου μπορούν να βοηθήσουν απευθεία στο διεθνές εμπόριο. Οι δυνατότητες του ψηφιακού εμπορίου ξεκινούν από το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι πλέον παγκόσμιο. 3,2 δι άνθρωποι βρίσκονται συνδεδεμένοι διαδικτυακά και ε, περίπου το 90% των ε, χωρών των ανθρώπων αυτών είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες και φυσικά πρέπει να υπάρχει και ε, δράση προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Νοέμβριο πέρσι για πρώτη φορά είχαμε περισσότερες κινητές συσκευέ στον κόσμο από ό,τι ανθρώπους και οι μισές από αυτές τις κινητές συσκευέ διαθέτουν και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 87% στον, αναπτυγμένο κόσμο και μόνο 40% στον αναπτυσσόμενο κόσμο και πριν από 5 χρόνια ήταν 5% η πρόσβαση σε κινητές συσκευές. Επομένως είναι τεράστια ανάπτυξη. Η πρόσβαση σε κινητές συσκευές ε, ενίσχυσε και τη δυνατότητα των κινητών εφαρμογών. Στην Ευρώπη μόνο ε, πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές και αυτό δημιουργεί και 400.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ε, υπάρχουν εφαρμογές που αφορούν ε, την κίνηση, τη ρήπανση, ε, υγεία, αθλητισμό. Για παράδειγμα, υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται DIS που βοηθά τα παιδιά με δυσλεξία και στέλνει τα στοιχεία σε ερευνητές στο πανεπιστήμιο που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βοηθήσουν. Υπάρχει μια Ιρλανδική εφαρμογή που βοηθά τα άτομα με δυσκολίες στην ε, στην ομιλία και το Angry Birds, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι μια εφαρμογή που ξεκίνησε από τη Φιλανδία και βοηθά τους ανθρώπους με την κατάθλιψη και το άγχος τους. Ε, διατίθεται σε πάρα πολλές γλώσσες δε. Τα ωφέλη για την παραγωγικότητα βοήθησαν το ΑΕΠ ε, των ΗΠΑ κατά 3,5%. Μεταξύ του 2003 και το 2010 περίπου το 17% της παραγωγικότητας στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό φυσικά μπορεί να αυξηθεί με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι ίσως πρόσβαση σε τεχνολογίες εχμής ε, οι οποίες είναι φθηνότερες διαδικτυακά. Είτε πρόκειται για cloud computer, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ε, δυνατότητες επικοινωνίες, το Skype, το WhatsApp, το Google Hangouts, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν, καθώς σε πρόσβαση σε δωρεάν ε, ε, πληροφορίες marketing, που θεωρείται ότι είναι ένας από τους βασικούς φραγμούς που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται παγκοσμίω. Επίσης, υπάρχει μια άλλη αναπτυσσόμενη αγορά που μέχρι το 2030 αναμένεται να έχει κύκλο εργασιών πάνω από 300 δισεκατομμύρια ε, εκατομμύρια ευρώ. Χρησιμοποιούνται ραδιοφωνικές συχνότητες ήδη από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για να βελτιώσουν κατά 15% την ε, ροή δεδομένων. Και αυτό δείχνει και πόσο σημαντικά είναι τα big data. Το ίντερνετ των πραγμάτων ε, βοηθά τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις παγκοσμίω, αλλά και οι άνθρωποι να συλλέγουν πληροφορίες για να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν την παραγωγικότητα. Και αυτά φυσικά δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις, βοηθούν και την ανθρώπινη υγεία και τις κυβερνητικέ. Ε, Δείτε για παράδειγμα ε, κατά τη διάρκεια του τυφώνα στις Φιλιππίνες τι συνέβη. Ε, υπήρχαν ε, υπηρεσίες κατεπίγουσας ανάγκης εκεί που χρειάζονταν χάρη στο διαδίκτυο και τα big data θα είναι το μέλλον της καινοτομία και της παραγωγικότητας. Τέλος, οι αλυσίδες διανομής δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν παγκοσμίως τα big data. Για παράδειγμα, υπάρχει μια φιλανδική επιχείρηση που χρησιμοποιεί τα big data, τα αναλύει στη Δανία για να δει τις διαφορές της θερμοκρασίας, την ταχύτητα του ανέμου και όλα αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να δούμε ε, πότε μπορεί να χρειάζεται αλλαγή σε εξαρτήματα, σε αποθήκες οι οποίες μπορεί να είναι στην Ασία και να σταλούν ε, ανταλλακτικά σε μια επιχείρηση στην Αυστραλία πριν υπάρχουν προβλήματα. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και επηρεάζουν τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο. Μέσω των διαδικτυακών αυτών ε, δομών από τις πλατφόρμες αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται παγκοσμίω. Το 90% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ ε, στο eBay μπορούν να κάνουν εξαγωγέ και αυτό φυσικά βοηθάει πολύ περισσότερο από το συμβατικό τρόπος. Ένα 12% μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάνουν ψηφιακό εμπόριο, ε, το 90% των ε, το 93% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο eBay έχουν και εξαγωγέ στο εξωτερικό. Επίση, επηρεάζουν τη σύνθεση του διεθνού εμπορίου και τη δυνατότητα να γίνεται εμπόριο σε υπηρεσίε και αγαθά χαμηλή αξία. Ε, δείτε για παράδειγμα την πρόσβαση σε υπηρεσίες που αναφέραμε, υγεία, παιδεία, το ψηφιακό εμπόριο επίσης ανθεί ε, και θολώνει τη διαφορά μεταξύ ε, υπηρεσιών που ε, ήταν διαθέσιμες ως φυσικά αγαθά στο παρελθόν. Τώρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να αγοράσει βιβλία, μουσική κλπ. μέσω διαδικτύου. Η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων ε, σε, ε, στο διεθνές εμπόριο είναι πάρα πολύ πιο εύκολη τώρα. Πολύ συχνά προσφέρουν ε, προϊόντα χαμηλής αξίας, πολύ απλά αγαθά, ενώ στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ ακριβά τα αγαθά που μπορούσαν να προσφερθούν διεθνώς. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον και εδώ έρχομαι να ενισχύσω και σε αυτό που είπε ο Ριουπέρτ ότι ένα από τα βασικά στοιχεία είναι να διασφαλέσουμε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο διαδικτυακό εμπόριο. Ε, είτε πρόκειται για εμπιστοσύνη για τα προσωπικά δεδομένα που δίνει κάποιο στη διάρκεια μια εμπορική συναλλαγή ε, και το κατά πόσο προστατεύονται, όπω επίση προστασία των καταναλωτών από ψευδεί πρακτικέ και να μπορεί να επιληθεί μια διαφορά εγκαίρω και με αποτελεσματικό τρόπο και φυσικά να είναι ε, εύκολη και ασφαλή η πρόσβαση. Ορισμένοι από τους φραγμούς στο ψηφιακό εμπόριο είναι από τους παλιούς ε, φραγμούς, αλλά γίνονται πιο σημαντικοί. Για παράδειγμα, τελωνιακές διαδικασίες, εφαρμογή για τον ε, κανόνα του, ίσονου ίσονους δασμού. Ε, και τέλος, ε, το διαδίκτυο και η δυνατότητα να δίνονται δεδομένα παγκοσμίω πρέπει να γίνεται δωρεάν. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί να είναι προβληματική η πρόσβαση στο διαδόκτυο. Καταρχάς, αυξάνεται το κόστος πρόσβασης στις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στο cloud computing, και κάποιες χώρες, κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεν έχουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση. Γι' αυτό και κάποιες επιχειρήσεις απλώς κάμπτουν αυτές τις αγορές ε, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ο αναπτυσσόμενο κόσμο λοιπόν θα πληγεί περισσότερο αν δεν αρθούν οι φραγμοί. Η Κίνα, η Ρώσα και η Ινδία έχουν προτείνει να έχουν διαφορετικού τρόπου ε, ε, νομοθεσία για τα δεδομένα αυτά και το που βρίσκονται. Ε, θα πρέπει να μπορούν να δίνονται δεδομένα πολύ εύκολα και θα υπάρχουν βέβαια και κάποιοι θέματα όσον αφορά τα ρυθμιστικά ζητήματα, είτε είναι η προστασία των καταναλωτών, η υγεία, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν οι θύνοντες να βελτιώσουν τις δυνατότητες να παρέχουν ε, υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη πρόσβαση υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. Πρέπει να διευκολύνουμε λοιπόν την ε, διασυνοριακή συνεργασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν κάλλιστα να προσφέρουν κατόλους κανόνες ώστε να έχουμε ένα παγκόσμιο διαδίκτυο και εδώ η διαλειτουργικότητα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δημιουργεί γέφυρες ε, μεταξύ των ηθινόντων και του κοινού. Ε, Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, και μπορούν να παραβιαστούν ε, το πρόσφατο περιστατικό ιδιωτικότητας ε, των δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ είναι σαφές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχουν ε, συγκεκριμένε εξαιρέσει για τα πνευματικά δικαιώματα και οι ευθύνε και αυτέ ήταν πάρα πολύ σημαντικέ ε, για την ανάπτυξη των ψηφιακών επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα κατάλληλο πλαίσιο για ρυθμιστική συνεργασία και να βελτιώσουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο διαδίκτυο και στι ροέ δεδομένων. Η πρόσφατη συμφωνία ε, με τις χώρες του Ειρηνικού και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Trans-Pacific, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία ε, βοηθούν σε συνεργασία για τα ψηφιακά ζητήματα και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις εκεί. Ε, υπάρχουν λοιπόν συμφωνίες επίσης υποδιαπραγμάτευση όπως η TIPT που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εδώ. Υπάρχει επίσης και ένα ενδιαφέρον για να κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο ΠΟΕ για το ψηφιακό εμπόριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα εσείς έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό καθένας. Ο κύριος Φύσας έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις παρεμβάσεις σας, οι οποίες μου φαίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ε, και εγώ ε, συμμετέχω και στην Επιτροπή Πολιτισμού. Και στην Επιτροπή Πολιτισμού υπάρχουν δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν πολύ συγκεκριμένα. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε, την προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, το copyright. Πώς μπορεί να γίνεται αποτελεσματική προστασία και με καλό τρόπο και επίσης ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο φορά τις εξαγωγές, ε, τις παράνομες συναλλαγές που γίνονται μέσω διαδικτύου ε, και στον αθλητισμό. είναι, αυτό είναι το βασικό καρκίνωμα του αθλητισμού και δεν υπάρχει κάποια λύση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα εσείς προκειμένου να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μακουλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη δημόσια κρόση, να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι ο ρυθμός με τον οποίο διαπραγματευόμαστε διεθνείς συμφωνίες είναι πολύ πιο ταχύς από την εξέλιξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς προσπαθούμε να άρουμε τους ε, ε υφιστάμενους ε, ε, φραγμούς για τις 28 χώρες ε, μέλη και ε, φραγμούς για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα στοιχείο το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ δύσκολα θα εξελιχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο αν δεν δώσουμε κατάλληλες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες πέραν των κατάλληλων υποδομών που επισήμανε ο πρώτος ομιλητής αλλά πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του ηλεκτρονικού εμπορίου και ε, όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, είναι πολύ σημαντικό και το είπαν και οι δύο ομιλητές ε, να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η νέα νομοθεσία, ενώ οι κανόνε μάλλον συγγνώμη, που χρειάζονται σε επίπεδο ΠΟΕ προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι νέε προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και με ποιο τρόπο ε, τα επεξεργάζεται τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για ε, τα θέματα του ΠΟΕ. Η κυρία Κερτών Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ και του δύο προσκεκλημένου. Δεν πιστεύω πως αμφιβάλλει κανεί για τι ευκαιρίε που δημιουργεί το διαδίκτυο και το δυναμικό επίση για τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Ε, στο Σάντερλαντ, την περιοχή από όπου κατάγομαι, τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία χρησιμοποιούνται για καινοτόμε δράσει, για να χτίσουν πάνω στο ψηφιακό κεφάλαιο. Κάτι το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτέ τι ευκαιρίε που αναφέρατε και στηρίζει θέσει ε, εργασία στην περιοχή. Προσπαθώ λοιπόν να πλαισιώσω με αυτόν τον τρόπο την ερώτησή μου. Σίγουρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, όμω όπω είπε και εσύ, Ρουπέρτε, υπάρχουν μεγάλε ανησυχίε για την ιδιωτικότητα. Και, η, οργανισμό, ένας οργανισμός καταναλωτών τοποθετήθηκε πάνω στι ανησυχίε αυτέ, επιχειρηματολογώντα ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και χρηματοπιστωτικέ ε, υπηρεσίε και τα αντίστοιχα κεφάλαια δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώ την ιδιωτικότητα. Εσεί λοιπόν τι έχετε να πείτε για την κριτική αυτή που ασκήθηκε στι υφιστάμενε εμπορικέ συμφωνίε. Ξέρω πώ έχει απαντήσει για το τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με τη συμφωνία ΤΙΖΑ, όμως η συμφωνία ε, ΣΕΤΑ έχει ολοκληρωθεί και τι λοιπόν να πεις γι' αυτό. Ε, κυρία Ρέντιν έχει το λόγο. Τρεις ερωτήσεις έχω εγώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, όταν μιλάμε για ψηφιακές ε, υπηρεσίες, ε, Ξέρουμε τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του. Δηλαδή μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, να επανακατασταθούν στο εξωτερικό για να αποφύγουν φορολογία για παράδειγμα. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό καθεστώς προστασίας όπως για, εκείνο για τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες. Έπειτα τα κεφάλαια και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες πρότυπες ρήτρε, όπως για παράδειγμα στο χώρο του ICS και τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές οι ρήτρε. Η προλαλή σας ήδη αναφέρθηκε σε αυτά τα προβλήματα πρέπει να περιλαμβάνεται η ελεύθερη ροή δεδομένων, να προλαμβάνεται η αναγκαστική προσαρμογή κατά τόπους, να, ε, να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία και να υπάρχουν και κάποιες γενικές εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα θέματα εθνικής ασφάλειας και να τηρείται φυσικά η αρχή της αναλογικότητας και τα κριτήρια της αναλογικότητας. Και αυτό με φέρνει στην επόμενη ερώτηση. Το άρθρο 14 σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Είναι, ε, καλύπτει τα πάντα ή πρέπει να ανατρέξουμε σε άλλα άρθρα, όπως για παράδειγμα στη Συμφωνία TPP, όπου αυτό το κείμενο έχει αντικατασταθεί με αναφορές στην αναλογικότητα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίτια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για αυτήν την ακρόαση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις ευρύτερες επιπτώσεις, διότι βλέπουμε ολόνα και περισσότερες εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτές οι εξελίξεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα από την πολιτική που εμείς χαράσουμε. Και πιστεύω πως πραγματικά αποτελεί πρόκληση αυτό. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Σλέγγελ Μίλχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε αρκετέ προτάσεις αύριο σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά και αναρωτιέμαι κατά πόσο θεωρείτε ότι το εμπόριο έχει ενσωματωθεί στις προτάσεις αυτές για την ψηφιακή αγορά. Αναφερθήκατε εν συντομία στη, στην εσωτερική αγορά, σε αντιδιαστολή με την ενιαία αγορά, όμως μου φαίνεται πως δεν υπάρχουν σαφή όρια, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρότυπα για παράδειγμα ε, την ασφάλεια ή την προστασία δεδομένων ή την ε, ευθύνη στο ε, διαδίκτυο στις εμπορικές συναλλαγές. Επίσης, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, αναρωτιέμαι κατά πόσο το εμπόριο και η μέση διάταξη για το εμπόριο συνδέονται με την εμπορική ατζέντα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ή όποιου είναι αρμόδιος τέλος πάντων και πόσο αυτές μπορούν να συνδυαστούν. Έπειτα, ε, η κυρία Ρέντινγκ μας ε, μίλησε για τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια και, την προστα... και τις προσωπικές ελευθερίες των χρηστών στο διαδίκτυο. Έπειτα, ε, η, η αναγκαστική προσαρμογή κατά τόπους και οι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ ακούω αρκετέ ε, κατηγορίε κυρίως από τι Ηνωμένε Πολιτείε που κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για προστατευτισμό, κατηγορούν τους Ευρωπαίους πολίτε ότι είναι υπερευαίσθητοι για τα προσωπικά τους ε, δικαιώματα και την προσωπική ε, πνευματική ιδιοκτησία τους. Ακούω ότι υπάρχει κλονισμός εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα από τους χρήστες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους προσκεκλημένους αν έχουν κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία έτσι ώστε να αποτρέψουμε την ε, αναγκαστική προσαρμογή κατά τόπους σε ορισμένα πολιταρχικά καθεστώτα και να οδηγηθούμε προς ε, ανοιχτές οικονομίες, κάτι που πιστεύω θα ωφελήσει όλους. Ευχαριστώ πολύ, ο Χέλμου Τσόλιτς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία δημοσίευση για την διακυβέρνηση στο διαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρει λοιπόν αυτή η δημοσίευση ότι ε, όταν ε, συνα... γίνονται συναλλαγές στο ε, διαδίκτυο λειτουργούμε καλή την πίστη και βάσει εμπιστοσύνη. Οι ροές δεδομένων είναι ανοιχτές σε όλους αλλά υπάρχει επίσης και ένα νομικό πλαίσιο ε, μέσα στο οποίο πρέπει να γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Όταν λοιπόν γίνεται λόγος για τις ε, προκλήσεις και τα βασικά στοιχεία της ψηφιακής αγοράς και το πώς θα αναπτύξουμε δυνατότητες, πρέπει να μην χάνουμε αυτό, το, αυτή τη σημαντική πτυχή. Διαβάζουμε το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό αναφέρει 400 εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτήν την συνεργασία, σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Πώς λοιπόν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις προκλήσεις με τη διασφάλιση ότι θα καλύπτονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε και ο κύριος Πώς μπορούμε δηλαδή να ε, ισχυριζόμαστε ότι αυτή η εμπιστοσύνη είναι και παράγοντα σταθεροποίηση. Μετά, πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ροή δεδομένων. Αν υπάρχει αυτή η ελευθερία στη ροή, όπως είπε και ο κύριος Λέγκελμιλ, τι σημαίνει δηλαδή στην ουσία. Σίγουρα αυτή η ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να συνεχίσουμε το καλό έργο Συμφωνείτε κι εσείς κύριε Πρόεδρε. Θα, συμφωνεί, θα σταματήσω όμως εδώ ε, για να μην υπερβώ το χρονικό όριο του ενός λεπτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, το δεύτερο σκέλος αφορά το άλλο πάνελ, όμως τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σλέγγελμιλ για τρία λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ε, ήταν όλες εύστοχες και τις επό... τους επόμενους μήνες και χρόνια θα πρέπει να προσέξουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Η κατάχρηση του διαδικτύου με τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα δεν είναι άμεσα θέμα του, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, αλλά παρόλα αυτά εντάσσεται σε αυτό το τομέα, αλλά ε, σχετίζεται περισσότερο με την ε, αστυνομία, το ίδιο με την αστυνομική δράση, όπως και η πορνογραφία παραδείγματος χάρη. Είναι πραγματική πρόκληση και το εξετάζουμε με τα κράτη-μέλη, αλλά είναι θέμα ε, επιβολής του νόμου. Δεν μπορώ σε αυτή τη χρονική στιγμή, όταν μιλάμε και εξετάζουμε το δυναμικό τη ψηφιακή οικονομία να δώσω πιο συγκεκριμένες απαντήσει. Ε, κύριε Ροντρίκε, ε, σε ποιο σημείο είμαστε, μα ρωτήσατε για την προσέγγιση που υιοθετούμε σε σχέση με τον ΠΟΕ και η σχέση ανάμεσα σε εσωτερικέ και εξωτερικές ε, πολιτικές. Είναι διαρκή η πρόκληση και το είπατε, διότι είναι παγκόσμια η αγορά. Η ψηφιακή αγορά είναι παγκόσμια. Δεν είναι άμεσα θέμα αρμοδιότητας μου, οπότε δεν θα το σχολιάσω. Ε, έχουμε εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, είναι καταπληκτικοί οι κανόνες μας, όμως αυτά που ε, επιδιώκουμε στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να συνάδουν με αυτά που εφαρμόζουμε εσωτερικά και σίγουρα δεν θέλουμε να υπάρχουν συγκρούσεις ως προς την νομοθεσία προστασία των ιδιωτικών δομένων και των εξωτερικών ε, διατάξεων. Όπως είπε και η κυρία Ρέντινγκ, θα επανέλθω σε αυτό. Ας ε, επανέλθουμε στα βασικά. Έχουμε ε, και ας με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι του ΠΟΕ, τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουμε αναθεωρήσει αυτή τη βασική νομοθεσία και στο σενάριο μετά τον Αϊρόμπι αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς μπορούμε να δώσουμε μια νέα πνοή σε αυτές τις ε, νομοθετικές διατάξεις. Είναι απαραίτητο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και κάτι άλλο. Έχουμε τη ΣΥΤΑ, ε, τη συμφωνία με τον Καναδά και νομίζω ότι είναι θετικέ οι διατάξει ε, για την. Ε, ρωτήσατε, κυρία Ρέντινγκ, αν επαρκεί το άρθρο 14. Είναι η βασική προστασία στην κάτσε για την εμπορική πολιτική. Καλό είναι το άρθρο, αλλά δεν είναι και πολύ ειδικό. Και μην ξεχνάμε τις, τα δεδομένα θέσεις στο localization. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αγγίζει καν ο ΠΟΕ και θα πρέπει να δούμε την ισορροπία ανάμεσα στις ε, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Τι ε, μπορούμε να αιτιολογήσουμε, διότι υπάρχει το θέμα της σχέσης ΕΕ και ΕΠΑ και όλοι έχουμε απαιτήσει σε σχέση με τα δεδομένα θέσεις και όλοι χρειάζονται τέτοια δεδομένα, κυρίως οι υπηρεσίες ασφαλείας, πληροφοριών, ε, θέλουν να διατηρούν αυτά τα δεδομένα. Αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή δεν είναι ε, ελεύθερη η κυκλοφορία των δεδομένων χωρίς κανένα δεδομένο θέση. Το θέμα είναι να βρούμε μια ισορροπία, δηλαδή να μην περάσουμε στο πεδίο του προστατευτισμού γιατί θα είναι δυσανάλογα υψηλές οι απαιτήσει μας. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Δηλαδή αναλογικότητα είναι η απάντηση. Πέραν αυτού θα πρέπει να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε σχέση και με την Κάτσε. Βλέπω ότι αναβοσβήνει το φωτάκι, οπότε ίσως να σταματήσω εδώ. Πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα και να εμβαθύνουμε ίσως στο διάλογό μας ε, την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε. Κύριο Πολμέλτσε, εξαιρετικέ ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποιε. Ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ διαφορετικό η θέση σε σχέση με το παρελθόν, γιατί έχει ανοίξει το εμπόριο και θέλουμε να αναπτύξουμε κανόνε τόσο ώστε να διατηρήσουμε αυτό το άνοιγμα και όπου χρειαστεί να προστατευτούμε κατά την εισαγωγή μέτρων που να αποδειχθούν προβληματικά. Ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ ε, δεν είναι ότι είναι ένα περιβάλλον χωρίς κανόνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες στον ΠΟΕ που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμοι διότι στηρίζουν τις δυνατότητες ε, ε, του ψηφιακού εμπορίου για τις τηλεπικοινωνίες. Η ΓΚΑΤΣ, παραδείγματο χάρη, η προληπτική αρχή που εφαρμόζεται σε αυτές τις συμφωνίες μας βοηθά να εφαρμόζουμε αυτές τις δεσμεύσεις και έχει ουδέτερες επιπτώσεις ως προς την προσφορά υπηρεσιών. Δηλαδή, αν αναλάβατε δέσμευση ΓΚΑΤΣ ένα συγκεκριμένο τομέα. Αν τελικά μπορείτε να την εφαρμόσετε και επιγραμμικά, τότε δεν έχει ε, ε, καμία επίπτωση στην δέσμευση, όμω δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτό γιατί δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν την TTIP και την ΤΙΣΑ και ε, αυτές οι νέες συμφωνίες μπορούν να μα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πρόοδο και σε αυτό το τομέα είναι σε πολύ καλή θέση η και η ΕΕ για να αναπτύξουν ένα νέο, ε, κανονιστή, μια νέα κανονιστική δομή που μπορεί να λειτουργήσει ως μορφότυπος ε, αν έχει θετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, η κανονιστική πρόκληση ποιοτικά είναι διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν ή με τα προϊόντα. Παραδείγματο χάρη είχαμε τους δασμούς ε, στα σύνορα και μετά μας ανησυχούσαν, μας ανησυχούσαν συγγνώμη, οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Τώρα στην ψηφιακή οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα τα διασυνοριακά εμπόδια, ώστε να έχουν την εμπιστοσύνη οι κυβερνήσεις σε σχέση με την πρόσβαση ε, που χορηγείται στα σύνορα. Είναι το αντίστροφο και γι' αυτό σας μιλούσα για τις εξτernalities, τις ε, εξωτερικές πολιτικές μας, ε, διότι θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο πρώτα να αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Δεν σταματάνε τα δεδομένα στα σύνορα και το ξέρουμε όλοι και πιστεύω ότι σε, μια διατλαντική, σε ένα διατλαντικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο στη συνέχεια θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα στον ΠΟΕ πραγματεύονται το ζήτημα, αλλά όχι μόνο, ίσως σε άλλα φόρα κανονιστική συνεργασία, σε, σε πιο πλευρή βάση θα μπορούσαμε να φροντίσουμε ε, να καταλήξουμε στις απαραίτητες τελικά εμπορικές δεσμεύσεις. Α, ε, εντάχει. Θα, ήθελα να μιλήσω για τα θέματα διακυβέρνηση. Μία παρατήρηση να κάνω. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ διακριτές κοινότητε και όσο προχωράμε αυτό που δεν είναι σημαντικό είναι να φροντίσουμε να είναι καλό ο διάλογο ανάμεσα στι δύο διότι είναι δύο διαφορετικά πεδία ε, διακυβέρνηση ε, και είναι πολυμερέ αυτό το σύστημα διαχείριση. Δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που διεξάγονται οι εμπορικές ε, συναλλαγές, διαπραγματεύσει συγγνώμη, στα πλαίσια του ΠΟΕ και μην ξεχνάμε ότι το θέμα της ε, διακυβέρνησης ε, συνδέεται και με οικονομικά ζητήματα και εννοώ ότι θα πρέπει αυτές οι δύο κοινότητες, ο διάλογός τους θα πρέπει να ενισχυθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Θα συζητήσουμε λοιπόν τώρα τους ε, κανόνες, ε, σαφείς και διάφανοι κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο. Έχουμε εδώ τους εμπειρογνωμονές μας και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Τζον Higgins, Γενικό Διευθυντή του Digital Europe, για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που διοργανώσατε ε, μια πολύ κατάλληλη συνεδρίαση και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα από πλευράς Digital Europe να κάνουμε και εμείς κάποιες παρατηρήσεις. Η Digital Europe είναι μια οργάνωση που ε, εκπροσωπεί τον τεχνολογικό τομέα που προσφέρει αξία στην οικονομία και στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στην ιδιότητά μου μπορώ να έρθω σε επαφή με πραγματικά πολύ ωραίους ανθρώπους ε, πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στην Πρατισλάβα με τον πρόεδρο της Ένωση στη Σλοβακία. Είναι ένας ε, από τους παγκόσμιους ηγέτες ε, στο αυτοματοποιημένα οικιακά προϊόντα. Πολλά προϊόντα τα οποία βλέπουμε σήμερα στο ίντερνετ των πραγμάτων των καταναλωτών. ένα άλλο παράδειγμα ένα συνήθιστο παράδειγμα της συνέπειας που έχει η τεχνολογία στο ψηφιακό εμπόριο είναι ένα μέλος μας που ε, είναι στη Σόφια, στη Βουλγαρία και έχει μια επιχείρηση λογισμικού που κάνει προσωμείωση ε, ε, της ζωής σε ένα πλοίο που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια. Ε, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που βρίσκονται επί του σκάφους ε, να μην ε, πέφτουν στη θάλασσα εμπορευματοκιβώτια και να μπορούν να σώσουν τη ζωή τους, να μπορούν να κυκλοφορήσουν ανάμεσα στα ψηφιακά καλώδια που υπάρχουν σε αυτά τα, τα, τα πλοία. Ε, ήθελα να πω δύο λόγια για την άποψή μας για το ψηφιακό εμπόριο, αλλά ο Ρούπερ τα είπε τόσο καλά που δεν χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειες, διότι νομίζω ότι περιέγραψε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Θα σας δώσω μερικά προσωπικά παραδείγματα του τι σημαίνει για μένα. Εγώ στη δεκαετία του 90 μια επιχείρηση στο Σάντα Φέ, στο Νιου Μέξικο και στο Λονδίνο. Είχαμε δύο έδρες και οι μουσικοί μπορούσαν να παίξουν μαζί στο διαδίκτυο. Ήταν ένα ε, στούντιο ηχογραφήσεων ε, ε, το οποίο ήταν ψηφιακό. Και έτσι δεν χρειαζόταν να πηγαίνουμε στους μουσικούς επιτόπου που είχαμε μουσικούς από όλο τον κόσμο και μπορούσαν να δημιουργήσουν σε αυτό το virtual studio ηχογραφήσεων που είχαμε. Έτσι μπορούσαμε να έχουμε μια επικοινωνία και υπήρχε ένα είδους ψηφιακό εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα είχα το προνόμιο να προσδεύω ε, σε ένα φόρουμ ε, στρατηγικής πολιτικής ε, για την επιχειρηματικότητα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο συνέβη στην Καλιφέρμηνια στο κλάδο της μουσικής είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν θα είχα προβλέψει να είναι αντίστοιχα ενδιαφέρον και το στρατηγικό φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο εξετάσαμε λοιπόν σε αυτό το φόρουμ πολιτικής ήταν οι δυνατότητες που έχει η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί την ψηφιακή τεχνολογία και κυρίως αυτό αφορά την εσωτερική αγορά στην ε, ψηφιακή εποχή. Ε, διαπιστώσαμε ότι το 75% της ψηφιακής τεχνολογίας ε, στην Ευρώπη ε, προήλθε από τη χρήση ε, της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορία αυτή με, πήγε στο ανώβερο με τον Επίτροπο Ότιγκερ και τον αντίστοιχο εταίρο του από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως συντονιστή σε ένα πάνελ για τις διατλαντικές πτυχές της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Και δύο πράγματα με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα από εκείνη την εμπειρία. Το ένα είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, συμμετείχαν σε αυτό το πάνελ, που ήταν από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όπως ε, θεωρώ, είχαμε τη ΣΑΠ, τη Schneider Electric, μια γερμανική, ε, γαλλική ε, επιχείρηση. Είχαμε τη General Electric, την Bosch ε, και το λογισμικό της και είχαμε λοιπόν επιχειρήσει από τις δύο πλευρές του ε, Ατλαντικού. Αλλά ένας από τους πανελίστε, όταν αναφέρεστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προσπαθούσε να καταλάβω τι εννοείτε. Γιατί εννοούσατε τη Γρυλανδία, γιατί εμείς δεν βλέπουμε πια τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε ότι η αγορά μα είναι παγκόσμιε αγορέ. Και ένα άλλο ανέκδοτο το οποίο πραγματικά ε, με εξέπληξε είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο του βιομηχανικού διαδικτύου συστήθηκε μια οργάνωση πριν από κάνα δύο χρόνια για να μπορέσει να καθορίσει πρότυπα και προδιαγραφές στον τομέα αυτό και να υπάρχει και μια κοινή ε, γνώση το λέγαμε Industrial Internet Consortium. Πριν από δύο χρόνια δεν είχε κανένα μέλος. Πριν από ένα χρόνο είχε 100 επιχειρήσεις μέλη και τώρα έχει 255 μέλη επιχειρήσεις. Πριν από τρεις εβδομάδες ε, είναι αυτά τα στοιχεία, κατά πάσα πιθανότητα αυξήθηκαν. Ξεκίνησε στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά σήμερα είναι μειοψηφία επιχειρήσεις Ηνωμένων Πολιτειών, προεδρεύει Schneider Electric. Και εξετάζουν διάφορες ε, ε, περιπτώσεις ε, για το βιομηχανικό διαδίκτυο, περιπτώσεις όπως για παράδειγμα τη ροή δεδομένων ε, στο ίντερνετ των πραγμάτων, τον κόσμο του βιομηχανικού διαδικτύου, όπου αυτά τα δεδομένα περνούν πέραν των εθνικών συνόρων. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες του θέματος αυτού. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό το θέμα του διαδικτύου για το εμπόριο είναι στην πραγματικότητα εμπόριο στην ψηφιακή εποχή. Και είναι μία επέκταση αυτών που έκανα στο Φόρουμ Πολιτικής εγώ, που ήταν το εμπόριο στην ενιαία αγορά στην Ευρώπη, είναι το εμπόριο σε μια μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά στην ψηφιακή εποχή. Και νομίζω ότι αυτά που μας είπαν ο Ρούπερτ και ο κύριος Μέλτσερ, ουσιαστικά έφυξαν κάποια από τα θέματα τα οποία ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει όμως πράγματι να τα σκεφτούμε ως εμπόριο στην ψηφιακή εποχή εντός της ενίας αγοράς και από εκεί και πέρα ευρύτερα στην παγκόσμια κοινότητα. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν τα πράγματα και πρέπει να τα ξεσκεφτούμε όταν προσπαθούμε να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται. Νομίζω το πρώτο είναι κάτι το οποίο με εντυπωσίασε όταν ε, μίλησα στον Πασκάλ Λαμή για τις ε, σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες και μου εξήγησε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τις εμπορικές συμφωνίες ε, σήμερα σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονταν στο παρελθόν. Και μου εξήγησε ότι γίνεται αυτό διότι όταν αναφερόμαστε πλέον σε εμπορικές συμφωνίες δεν λέμε ότι αν μειώσετε εσείς λίγο τους δασμούς θα μειώσω και εγώ λίγο τους δικούς μας και γίνονται όλα αυτά και κλεισμένων των σειρών και γίνεται μια διαπραγμάτευση ε, με τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν είναι πια έτσι. Ε, πλέον έχουμε ρυθμιστική σύγκληση που μας ενδιαφέρει και αυτό φυσικά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον κόσμο ε, στον οποίο ζουν στις διάφορες πλευρές του κόσμου. Και το γεγονός ότι αφορά κυρίως νομοθετική σύγκληση σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη σημασία και είναι πιο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό ο κόσμος ενδιαφέρεται πλέον ε, για την νομοθεσία εκεί που ζει. Η άλλη σημαντική συνέπεια και νομίζω ότι προέκυψε και από κάποιες από τις ερωτήσεις ε, που ρώτησε και η κυρία Σχάκε αλλά και άλλοι και νομίζω ότι το ανέφερε και ο κύριος Μέτσλερ. Δεν μπορούμε αυτό το ψηφιακό εμπόριο να το εξετάσουμε μόνο υπό το πρίσμα του εμπορίου. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το ε, ψηφιακό εμπέριο έρχεται να διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε ε, τη σύγκληση σε νομοθετικό επίπεδο και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παγκοσμίω. Αλλάζει η προσέγγιση λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας και επομένως έχουμε δύο διακριτές κοινωνίες όταν αναφερόμαστε στο εμπόριο και στην διακυβέρνηση του διαδικτύου και όταν αναφερόμαστε σε παράνομα στοιχήματα, για παράδειγμα, στον αθλητισμό και πώς επηρεάζει αυτό τις εμπορικές συμφωνίες, ε, αρχίζουμε να εμπλέκουμε πάρα πολλές διαφορετικές κοινότητες και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο να το ε, γνωρίζουμε ως σημείο διαταραχής. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να βλέπουμε πλέον τα πάντα από το φακό του εμπορίου. Πρέπει να έρθουν να συμμετέχουν και οι άλλες κοινότητες που έχουν ενδιαφέρον είτε πρόκειται για κανόνες τηλεπικοινωνίες είτε για διακυβέρνηση του διαδικτύου είτε πρόκειται για παράνομα στοιχήματα αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να επιδείξει ευφυΐα, είναι να συγκεντρώσει αυτές τις διάφορες κοινότητες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι κάνουμε στην ενιαία ψηφιακή αγορά αντικατοπτρίζει και αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε στο ψηφιακό εμπόριο. Δεν ανταλλάσσουμε σημειώσεις, απλώς ε, ε, θα τους βλέπουμε ως ε, τμήμα του ίδιου μοσαϊκού. Και ένα τελευταίο και με το οποίο θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Ε, σε αυτό το νέο διαταραγμένο μοντέλο ε, στο οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε συνεργασία από τις διάφορες πτυχές της κοινότητας, είτε πρόκειται για διαπραγματευτές ε, σε επίπεδο εμπορίου, είτε ε, εμπειρογνώμονες σε θέματα διακυβέρνηση του διαδικτύου. Ο κλάδος του διαδικτύου είναι διατεθειμένος να βοηθήσει να βρούμε το δρόμο μέσα από όλα αυτά. Γιατί αυτό το που θέλουμε να επιτύχουμε εμείς είναι ο συνάδελφος ο οποίος ε, κάνει τη δουλειά του στη Σόφια στη Βουλγαρία δεν θα πρέπει να σκεφτεί καν το ψηφιακό εμπόριο, θα μπορεί να δραστηριοποιείται όπου θέλει, οπουδήποτε στον κόσμο και θα υπάρχουν κατάλληλοι εμπορικοί κανόνες για να τον υποστηρίξουν σε αυτό που θέλει να επιτύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα στο λόγο τον Ετζόκ Μακνάμι, εκτελεστικό διευθυντή της European Digital Rights. Έχετε το λόγο. Τζο Μακνάμι ονομάζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η European Digital Rights είναι μια ένωση που εξετάζει το διαδίκτυο από την άποψή του ότι είναι κάτι που μπορεί να ενισχύσει και να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για να συνεχίσω αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν από λίγο, ασχολούμαστε περισσότερο με το με την ψηφιακή τεχνολογία και το εμπόριο παρά με το ψηφιακό εμπόριο. Και προσπαθούμε να εξετάσουμε τις νέες ευκαιρίες που έχουμε στους χώρους αυτούς. Αναφέρθηκε η δυσκολία ε, στην ε, ταχύτητα αντίδραση της νομοθεσίας, στις ε, αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της τεχνολογίας. Και ίσως ένα μέρος της λύσης έχει να κάνει με τις αρχές που θα διέπουν την νομοθεσία. Γνωρίζουμε τις ευρωπαϊκές αρχές, ξέρουμε τι ε, περί πρόκειται. Και όταν η κυρία Ρέντινγκ άρχισε να ασχολείται με το θέμα, δεν άρχισε από το μηδέν, άρχισε με την οδηγία του 1995 που, ε, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες φυσικά ε, δεν είναι τόσο επίκαιρες αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα είναι πώς θα εξυγχρονιστούν αυτές οι αρχές. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επαναφεύρουμε την προσέγγιση μας και να επωφεληθούμε από τα αποτελέσματα. Κάτι ε, το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ακούγεται ε, πολύ και δρυμία κριτική στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι το έχουμε ακούσει φαντάζομαι. Όμως θα ήθελα εδώ να κάνουμε δύο βήματα πίσω και να ε, αναλογιστούμε το τι έχει γίνει σωστά. Και για να συνεχίσω σε αυτό που είπε ο κύριος Σλέγγελμιλ, στη δική του παρουσίαση ε, θα αναφερθώ στην ε, αγορά ε, τηλεπικοινωνιών. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση ψηφιακές τεχνολογίες χωρίς αυτό. Ο Τζόναθαν Χίλ, ο Επίτροπος από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρθηκε σε αυτό από τα, από τα πρώτα θέματα. Χρειαζόμαστε επιτυχία, να πάρουμε την επιτυχία των τηλεπικοινωνιών και να την μεταφέρουμε και μεταλαμπαδέσουμε στους άλλους τομείς κάθε Ευρωπαίος πολίτης πλέον έχει καλύτερες επιλογές, πιο οικονομικές επιλογές, χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Και εγώ προσωπικά είδα την εξέλιξη αυτή ε, με τα ίδια μου τα μάτια. Ε, είδα στο χωριό της Ιρλανδίας από το οποίο κατάγομαι οι επικοινωνίες να πηγαίνουν, ε, να γίνονται από μια μαύρη τρύπα, από μια κυρία στο ταχυδρομείο που ε, ε, ασκούσε καθήκοντα τηλεφωνήτρια ε, στο να έχει κάποιο μια μεγάλη ευρύτατη γκάμα επιλογών. Και η Ευρώπη ευθύνεται γι' αυτό. Η Ευρώπη το έκανε αυτό. Και το έκανε μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται στην συμφωνία αυτή ως ε, το εργαλείο που θα ανοίξει τις αγορές μας και στο εξωτερικό. Ε, πρέπει να διδαχθούμε από τις θετικές μας εμπειρίες, να ε, χρησιμοποιήσουμε τους κανονισμούς για να μας βοηθήσουν και στο μέλλον. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και βλέπουμε και ότι υπάρχει μία τάση για υπερβολική νομοθεσία. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μας ε, δείχνουν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να πιέσουν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επίσης βλέπουμε ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών τίνει να ενοποιείται για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφύγουμε αυτό ακριβώς ακούστηκε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει ε, και τις επιχειρήσεις. Όχι, πρέπει να οδηγηθούμε σε μια νομοθεσία η οποία θα επιφέρει ε, δίκαιες πρακτικές και γι' αυτό χρειάζεται να διασφαλίσουμε ε, τη συνέχεια αυτής της επιτυχίας που είχαμε σε άλλους τομείς. Διότι η Ευρώπη το χρωστά αυτό στους πολίτες της, να συνεχίζει να προσπαθεί για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία, ε, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως είπα και πριν, μόλις έγινε μια αναθεώρηση ε, των αρχών της ε, νομοθεσίας περί προσωπικής, προσωπικών δεδομένων, η οποία νομοθεσία αποτελεί βάση για αντίστοιχη νομοθεσία στον υπόλοιπο κόσμο. Και πρέπει να αποφύγουμε να αποδυναμωθούν τα πρότυπα προστασίας δεδομένων και αυτό κινδυνεύει να γίνει και να θυσιαστεί η προσωπική ζωή και ιδιωτικότητα στο βωμό της ανάπτυξης. Το επιχείρημα είναι λοιπόν ακριβώς αυτό. Και αυτή η τάση φαίνεται στην επιστολή 14 χρόνων στην Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία καλεί για την ε, ισορροπία ανάμεσα στα ψηφιακά προϊόντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία δεδομένων. Ε, δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα δύο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει επίσης να αποφύγουμε την ευελιξία στις εμπορικές συμφωνίες, η οποία θα ε, προκαλέσει πτώση πτώση ε, των ε, προτύπων, πτώση των συνθήκων. Και εδώ πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι εθνικές διοικήσεις, διότι αυτή τη στιγμή στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, το 45% των επιχειρήσεων έχει πει ότι η προστασία των δεδομένων τους έχει εμποδίσει στις συναλλαγές και έχει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Τώρα, οι ανησυχίε για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα απασχολούν ε, πολλούς, εκατομμύρια πολίτες ε, και οδηγούν σε ύφεση στις αγορές που θα έπρεπε να είναι το ακριβώς αντίθετο. ακούμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφίσει έναν οριζόντιο κανονισμό για την ψηφιακή εποχή που περιέχει προστασία προσωπικών δεδομένων ε, στις ψηφιακές ε, τεχνολογίες και έχει οδηγήσει στην άνθηση των ε, startup. Η επιτυχία αυτή είναι βασισμένη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ε, κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι και να μας δίνει όθεση να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Ε, τώρα, ο κανονισμός πιστεύω πως πρέπει να παραμείνει μια δημοκρατική απόφαση. Τα μέτρα που θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα ε, νομίζω έχουν ληφθεί μέτρα ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκαν 7 φορές που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο σχετικά, αλλά δεν νομίζω ότι τις μέτρες θα δεν βγαίνουν τόσες. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να υπερασπιζόμαστε αυτά τα δικαιώματα, διότι η αποτυχία μας να το κάνουμε θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην αγορά στο εξωτερικό. Οι ρήτρες και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας ΤΙΖΑ πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους. Τώρα, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδανική. Αναμένεται ακόμα η έγκριση, αλλά έχουν ήδη διατυπωθεί ορισμένε επιφυλάξεις στο σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο έχει υποβληθεί από τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το εμπόριο και την εσωτερική μας πολιτική. οι διαρροές που έχουν γίνει σχετικά με τις σχετικές με τον DSM προτάσεις είναι ανησυχητικές. Διότι βλέπουμε ένα πολύπλοκο καθεστώς ε, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να το διορθώσει. Ενδεχομένως να προτείνει κάποια πρόσθετα μέτρα για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας για να γίνει πιο δύσκολη η κλοπή όμως αυτή τη στιγμή εξετάζονται διάφορες διατάξεις, διάφορα εθελοντικά μέτρα που θα λαμβάνουν οι πάροχοι ίντερνετ. Όμως και οι πάροχοι και οι ε, διαφορετικές χώρες θέλουν άλλα πράγματα και εφαρμόζουν εθελοντικά αυτές τις ε, προτάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέοι φραγμοί από εκεί που δεν υπήρχαν και να διαπιστώνονται παραβιάσεις στην νομοθεσία. Επίσης, η αντιτρομοκρατική οδηγία δεν περιέχει εκτίμηση αντικτύπου και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει ο γεωγραφικός ε, αποκλεισμός, υπάρχει το κακόβουλο λογισμικό κρυπτογράφηση, για όλα αυτά δεν έχει γίνει εκτίμηση αντικτύπου, ούτε καν έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμηση αντικτύπου. Ελπίζω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει αυτό που είπε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, δηλαδή να υποβάλει προτάσεις που θα άρουν αυτούς τους φραγμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η Μαρίτια. Thank you, Chair. That was faster than... Ευχαριστώ. Δεν περίμενα να μου δώσετε το λόγο τόσο γρήγορα. Περίμενα πλήθος ερωτήσεων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρεμβάσεις και ζωτική σημασία για τη σημερινή μα συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι που φαίνεται προφανές, αλλά το εμπορικό ζήτημα θέλω να το βάλουμε στα γενικότερα συμφραζόμενα και απευθύνομαι και στου δύο μιλητές. Η εμπορική πολιτική, ποια σημασία έχει σε αυτό το πλαίσιο. Ο κύριος ε, Μακνάμι μα μίλησε ε, για την αναντίστοιχη ανάμεσα στις, ε, στην τεχνολογική πρόοδο και στην ε, εκπόνηση οποιασδήποτε πολιτική πολιτικής γενικότερα. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα μέτρα, ποιους άλλους τρόπους θα είχαμε για να ανοίξουμε το δρόμο για το ψηφιακό εμπόριο, για να ενισχύσουμε, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των χρηστών και των καταναλωτών επιγραμμικά, και να εφαρμόσουμε τις αρχές όπου ανέκαθεν είχε ηγετικό ρόλο η Ένωση. Ίσως και οι δύο μιλητές μπορούν να μας μιλήσουν για την παρακολούθηση του ανοιχτού ίντερνετ και την ε, μαζική λογοκρισία όχι μόνο ως προς ε, την ε, πλευρά του εμπορικού φραγμού αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την συγκρότηση κανονιστικού πλαισίου αφενός και αφετέρου της χρήσης των τεχνολογιών παγκοσμίως. Επίση, ε, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι εξαγωγικοί έλεγχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη μαζική παρακολούθηση, υποκλοπή κτλ που ε, ενδεχομένως μπορούν να πλήξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Αυτή η υπερσυνδεσιμότητα που διαπιστώνεται ευρέω ε, στην παγκόσμια οικονομία και χάρη στο ανοιχτό ίντερνετ ε, αντιτίθεται κάθεται στη νομοθεσία σε επίπεδο κρατών μελών ή σε πολυμερές επίπεδο ενώ χρειαζόμαστε παγκόσμια, παγκόσμιας εμβέλειας κανόνες. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Χρειαζόμαστε τέτοιου κανόνε. Και ποιο, πώ θα μπορούσαμε να του επιτύχουμε, όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και γενικότερα για την διακυβέρνηση στο διαδίκτυο ούτως ώστε με τα ανοιχτά πρότυπα και τα ανοιχτά δικαιώματα να ε, προστατεύουμε, ε, να υπάρχει προστασία αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να λειτουργήσει το εμπόριο. Ευχαριστούμε. Ο Χέλμουντ. Επικόντας τη τελευταία παρατήρηση της Μαρίτιε, ε, ε, σε σχέση δηλαδή με την ερώτηση αν χρειαζόμαστε κανόνες παγκόσμιας εμβέλειας. Κάτι γνώμη μου, φυσικά χρειαζόμαστε παγκόσμια προσέγγιση, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Τώρα ερώτηση ε, προς τους δύο μιλητές. Στις είπα υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή για τα θέματα εθνικής ασφάλειας που να εποπτεύει την ροή δεδομένων και όλα αυτά που τώρα συζητάμε. Είναι εμπορικός φραγμός αυτός, γιατί και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ελέγχουμε τις ροές, αλλά ελέγχουμε και τους ιδιώτες έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει το, κράτο, κράτος ή είναι θέμα ε, προσωπικών δεδομένων ή ε, είναι απλώς ένας εμπορικός φραγμός επειδή αυτό το θέμα συζητάμε. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι Παραπονιόμαστε σε κάποια κράτη-μέλη ότι παρακολουθούν τα, ε, τη, ροή δεδομένων και περιορίζουν ελεύθερη κυκλοφορία γιατί επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Αφενός και αφετέρου για τη δική μας ασφάλεια ε, θεσπίζουμε νέα δικαιώματα για το κράτος, για την εποπτεία. Ίσως εσείς, ε, άρα και ο κύριος Σλέγγεν Μέλχ θα μπορούσαν ε, να μας απαντήσουν πώς να διαχειριστούμε αυτή την αντίφαση, γιατί χρειάζεται μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και μια συνολική προσέγγιση. Ο κύριος Λάγκη, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Το κανονιστικό μας σύστημα βασίζεται Ε, στη διαδικασία που ακολουθούμε για τη συγκρότηση κανόνων και νομοθετικών διατάξεων. Για το ψηφιακό εμπόριο είναι ο πλέον ε, ενδεδειγμένος τρόπος, ε, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και την τεχνολογική πρόοδο, γιατί πάντοτε ουραγοί είμαστε ως προς την, τις τεχνολογικές εξελίξεις. θα προτείνατε για να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Κυρίως όταν μιλάμε για κανόνες σε, σε παγκόσμιο επίπεδο. So, thank you for those very and... Απλές οι ερωτήσεις. Joe will in a Ο Τζο, θα μας τα πει σε λίγο, αλλά προς το παρόν να πω κι εγώ ότι... Πέραν κάθε αμφιβολίας, ό,τι μέσο έχω στη διάθεσή μα ε, για να έχουμε παγκόσμια πρότυπα, να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο παγκόσμια πρότυπα και άλλο παγκόσμια νομοθεσία. Παγκόσμια πρότυπα μπορούμε να έχουμε σε ένα τομέα, αλλά μην προσπαθούμε να τα, διευρύνουμε, να τα επεκτείνουμε και σε άλλου τομεί. Ε, Παραδείγματο χάρη για τι κρατικές προμηθείες, ε, ε, συγγνώμη, για το μοντέλο που χρησιμοποιούμε για την διακυβέρνηση στο διαδίκτυο, ισχυρίζεται κάποιοι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ευρύτερα σε άλλους τομείς. Ε, εκεί θα πρέπει να δούμε για τα εμπορικά ζητήματα, όμως υπάρχει ε, αντίφαση σε σχέση με τα ατομικά μας δικαιώματα. Και θα το συνδέσω αυτό με αυτά που συμβαίνουν με το, σε σχέση με το Brexit. Ε, μία διάσταση του ζητήματος είναι τι γίνεται με την εθνική κυριαρχία θέλετε να συμμετάσχετε σε μαζικότερες προσπάθειες με περισσότερους ανθρώπους, τότε χρειάζεται ε, μια διαδικασία συλλογικότερη για τη λήψη αποφάσεων και περνάμε από το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στο διεθνές, στο παγκόσμιο κτλ. Τι πρέπει να συζητήσουμε, σε ποιο επίπεδο και ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η ουσία. Οπότε υπάρχουν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη και είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Δεν μπορούμε εύκολα να τα διαπραγματευτούμε. Ε, όμως κάποια άλλα Αντίθετα, μπορούμε, παραδείγματο χάρη, τι λέμε ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να έχει 12 παίκτε, γιατί έτσι μπορούμε να ε, ε, κερδίσουμε περισσότερου αγώνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμω, τι να κάνουμε, άμα παίζουμε με του άλλου Ευρωπαίου, θα πρέπει να έχουμε 11 στην ομάδα. Και, παρόλα αυτά, ε, ναι, το επίπεδο της Γερμανίας δεν πρόκειται να το φτάσουμε, το ξέρω. Λοιπόν, ε, για τη μαζική λογοκρισία, μαζική παρακολούθηση και τα λοιπά, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Η ΕΠΑ και ο ΙΕΜ φέρνουν ευθύνη για τη συγκρότηση, για τη θέσπιση παγκοσμίου ε, προτύπου. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι παραδοσιακή ευρωπαϊκή προσέγγιση, μαζική παρακολούθηση βασίζεται στους κανόνες που δέχεται η κοινωνία στην Ευρώπη. Όμως τώρα όλοι οδηγούμαστε προς ένα κοινό πρότυπο ανάμεσα είπα και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ακόμα, αλλά νομίζω υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρότυπο αλλά ε, ένα κοινό πρόσωπο που θα επιτρέπει και την παρακολούθηση είναι μεγάλο βήμα ε, αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Ε, χρειαζόμαστε κοινέ αξίε. Σε ποιο βαθμό επιτρέπουμε την παρακολούθηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και θα πρέπει να εθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ να καταλήξουν και να κωδικοποιήσουν ένα τέτοιο κοινό πρότυπο. Uh, και εγώ θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά. Όσον αφορά τις μαζικές παρακολουθήσεις, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, έχουν χάσει σε σεβασμό ε, των ίδιων των αξιών. Ε, οι αποκαλύψεις στις Ηνωμένε Πολιτείες οδήγησαν ε, στους ε, δικαστές να διαμαρτύρονται ότι συστηματικά τους παραπλανούν. Υπάρχει και η πράξη η νομοθετική πράξη Πίτσιτ, η οποία προσέλαβε νέα σημασία από τότε που τελείωσε η διαδικασία. Όλα αυτά δεν σέβονται τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι ο κατεξοχήν τρόπος με τον οποίο ε, γίνεται ε, αναλογικά ο περιορισμό των θεμελωδιών ε, ελευθεριών. Αντιστοίχως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σαφεί εξαιρεσει. Αν μου εξηγήσει κάποιος επακριβώς ε, τι είναι εξαίρεση εθνικής ασφαλείας, ε, να το δεκτώ, αλλά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εγκρίθηκε νομοθεσία γνωρίζοντα πλήρω ότι ήταν παράνομη και χρειάστηκαν 7 χρόνια ώστε μια κυβερνητική οργάνωση να προσφύγει στο δικαστήριο για να αναστρέψει την απόφαση. Η οδηγία PNR PNR ε, εγκρίθηκε πριν από μερικέ εβδομάδες. Υπάρχει και ε, γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα. Ε, δεν είναι λοιπόν... κάτι το οποίο σέβεται τις βασικές μας αρχές, ούτε και αυτό. Όσον αφορά τη λογοκρισία, Υπάρχουν σαφείς κανόνες στο άρθρο 52 της χάρτας ότι οποιοδήποτε περιορισμός πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητος, επομένως πρέπει να επιτυγχάνει ε, στόχους γενικού ενδιαφέροντος, αλλά υπάρχουν ε, πάρα πολλά παραδείγματα ε, blocking στο διαδίκτυο που δεν βασίζονται στην ομοθεσία και ποτέ δεν αναθεωρούνται ως προς την αναλογικότητά τους. Ε, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορους τρόπους ζητά από ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, να περιορίσουν, να διαγράψουν ε, ή να μπλοκάρουν περιεχόμενο ε, τυχαία. λέει ο Χάρντο ότι πρέπει να καθορίζονται οι περιορισμοί και να δικαιολογούνται αλλά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς περιορίζει ε, τα δικαιώματα των επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι προβλέψιμο αν είναι μεγάλη, μικρή επιχείρηση, αν είναι νομοθεσία. Ε, υπάρχει μια υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία νομίζω ότι δημοσιεύθηκε χθε. Κάποιο επέκρινε μια κατασκευαστική εταιρεία σε μια ιστοσελίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαγράφηκε το περιεχόμενο γιατί κάποιος ε, διαμαρτυρήθηκε λόγω ε, νομοθεσίας Ηνωμένων Πολιτειών περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, και σε λίγες εβδομάδες θα υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρητορία μίσους και με ποιους μιλάει με τη Microsoft, το Facebook και το Twitter. Έχουν οικονομίες κλίμακας, οι χώρες τους έχουν τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Τι κάνουμε εμείς ε, για τη λογοκρισία. Έχουμε τη χάρτα, έχουμε τη σύμβαση και υπάρχει και το «Αχ, σας παρακαλώ κάντε κάτι ώστε να μην χρειαστεί να νομοθετήσουμε». Δεν αρκούν αυτά. και ε, συντομία θα συμφωνήσω με το Τζον. Είναι πάρα πολύ καλό το μοντέλο. Είναι πολύ δύσκολο όμως να το πετύχουμε σωστά αυτό το μοντέλο. Η αρχή είναι σωστή να έχουμε τις κατάλληλες οργανώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις με την κατάλληλη πυρογνωμοσύνη και να είναι σταθμισμένα όλα αυτά κατά τρόπον ώστε να γίνονται σεβαστές και οι περιφέρειές τους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Ε, δεν είναι αυτό το συλλογικό μοντέλο ένα τέλειο πλήρες μοντέλο. Σίγουρα υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται η ακρόασή μας και για να είμαι ειλικρινής δεν έχουν απαντηθεί όλα με τα ερωτηματικά. Ίσως να είμαστε απλώς στην αρχή μιας διαδικασίας. Ε, προσπαθούμε να δούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές μας ε, για την πολύ σημαντική τους ε, συνεισφορά ε, σήμερα και τη συζήτηση και όλα αυτά θα τα έχουμε και σε συγκεκριμένες συμφωνίες εμπορίου. Ελπίζουμε και στην DTIP και σε άλλες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αυτό ολοκληρώνεται και η συνεδρία της Επιτροπής μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο υπό τα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση 15 και 16 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ.